Λοιπόν. Um, Κυρίε και κύριοι, λέει ο Πρόεδρο, Α αρχίσουμε την σημερινή μα συνεδρίαση. Δυστυχώ, ο κύριο Μωρά, ο προεδρό μα, δεν μπορούσε να παραστεί, οπότε έχω εγώ τη χαρά και το προνόμιο να προεδρεύσω για σήμερα. Το πρώτο μα θέμα είναι η έγκριση της ημερησίας διατάξεως. Υπάρχει μια αλλαγή. Σημειώσατε ότι το σημείο υπαριθμών 13 όσον αφορά τον ΦΠΑ και καταπολέμηση των σχετικών απατών αναβάλλεται και θα ζητήσει την επόμενη συνάντηση. Επομένως το 13 πάει για την επόμενη συνεδρίαση. Άρα δεν έχει ένσταση για την ημερησία άταξη όπως τροποποιήθηκε. Θεωρούμε ότι εγκρίνεται. Δεν υπάρχει αντίρρηση, επομένω εγκρίνεται. Επίση λάβετε υπόψη ότι δυστυχώ η διερμηνία προ τα και από τα κροατικά τέλο πάντων και κελτικά σήμερα δεν υπάρχει. Επίση, η έγκριση των προτάσεων και συστάσεων των συντονιστών Πρόκειται για τον ορισμό εισηγητών. Ο κύριος Μπόνι του ΕΛΚ, οριστική εισηγητής για την έκθεση Πρωτοβουλία που αφορά την Επιτροπή την νομική και ονομάζεται ε, το αστικό δίκαιο και η ρομποτική η κυρία Βίξτρομ της ε, Άλντε ορίστηκε η συγκήτρια για τα κριτήρια και μηχανισμούς που θα καθορίσουν τα αρμόδια κρατή μέλη για την εξέταση μιας αίτησης διεθνούς προστασίας η οποία αίτηση υποβάλλεται ε, σε κάποιο κράτος μέλος από κάποιον ε, πολίτη της χώρας ή από κάποιον απάτριδα. Επίσης, ο κύριος Κέρκοπ ορίστηκε για την Eurodac ε, εισηγητής. Συμφωνείτε με αυτέ τι προτάσει των συντονιστών. Ωραία, προχωρούμε τότε και πάμε στο πρώτο σημείο της μεσαίας διατάξεως. Υπάρχει 3 στη σειρά και μιλάμε για την δημιουργία της βάσης δεδομένων γύρω όσον αφορά τη σύγκριση των αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του σχετικού κανονισμού που αφορά την ε, ταυτοποίηση κάποιου παρανόμως ε, διαμένοντος ε, πολίτη τρίτης χώρας ή κάποιου απάτριδος. Ο κύριος Κέρκοπ είναι ο εισηγητής. Άρα πρώτα πρώτα έχουμε την εισήγηση της Επιτροπής. Στις 4 Μαΐου είχε κατεβάσει την οφειλής πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια μιας ευρείας μεταρρύθμισης του κοινού συστήματος ασύλου. σε σχέση και με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6 του 2016. Και είπαμε ότι αυτή η μεταρρύθμιση αφορά την μεταρρύθμιση του Δήμου του Δουβλίνου και επομένως και το γεροντάκι θα πρέπει να προσαρμοστεί και ο σκοπός είναι να επεκταθεί η ε, λειτουργία, ούτως ώστε να διευκολύνει τι επιστροφέ και αντιμετώπιση τη λαθρομετανάστευση Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επίση έχει υποβάλει μια πρόταση, ούτω ώστε να υπάρξει επαναξιολόγηση και μάλλον αναθεώρηση του κανονισμού της Eurodac. Θα παρουσιάσει ε, την ε, πρόταση ο τμήματάρχη τη γενική διεύθυνση των Ιστορικών Υποθέσεων και Ασύλου, ο κ. Και έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που δίνετε αυτή την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την πρότασή μας όσον αφορά τον κανονισμό για την Eurodac. Να σας πω με δύο λόγια ποια είναι τα βασικά σημεία, βασικές αλλαγές, τροποποίησης του ισχύοντος κανονισμού. Πρώτα-πρώτα, όπως αναφέρατε, Πρόεδρε, έχουμε κάποιες τροποποίησεις για να προσαρμοστεί η Eurodac αλλά και η εφαρμογή της στο σύστημα του Δουβλίνου, κάτι το οποίο προχωράει παράλληλα. Και επίσης θέλουμε να υπάρξει διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή ε, της ε, Eurodac για να καλύψει και την λαθρομετανάστευση. Να υπάρχει δηλαδή ε, αποθήκευση δεδομένων κάποιων πολιτών τρίτων χωρών που δεν έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου. Οπότε θέλουμε εδώ να έχουμε τη συγκρισιμότητα των στοιχείων του Eurodac. Φερρυπίν για κάποιον παρανόμως διαμένοντα θα γίνονται οι συγκρίσεις με αυτούς οι οποίοι διέβησαν παρανόμως στα εξωτερικά σύνορα. Επίσης είπαμε ότι θα πρέπει από τα 14 να κατέβει το όριο λήψη αποτυπωμάτων, να πάει από τα 14 ή στο 6. Να δούμε επομένω τι είναι πρακτικό και τι είναι εφικτό σε σχέση και με την ε, αποθήκευση των ε, ε, αποτυπωμάτων ανηλίκων και είπαμε να καλυφθούν από το σύστημα του Δουβλίνου. Και αυτοί οι ανήλικοι επίση είπαμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα εργαλείο τόσο στα κράτη-μέλη να μπορούν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν αγνοούμενου ανηλίκους. Όταν, ας πούμε, έχουμε κάποια οικογένεια, του Ντεσάσιλου έρχονται ε, και χωρίζουν τα παιδιά από του ε, γονεί βοηθά στο να ξαναβρούμε τα παιδιά και να γίνει πανένωση, το να έχουμε τα δακτυλικά αποτυπώματα. Επίση, μπορούν έτσι να παρακολουθήσουμε το τι έγινε με κάποιου ασυνόδου ανηλίκου που πολλέ φορέ ζητούν διεθνή προστασία και που φεύγουν από τα ε, κέντρα φιλοξενία. Οπότε και εδώ βοηθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα. Επίση, προτείνουμε σε κάποιε συγκεκριμένε ε, συνθήκε να αξιοποιούνται τα στοιχεία τη Eurodac για τους επαναπατρισμούς, τις επιστροφές, ε, συνεργασία με τις τρίτε χώρες. Ε, αυτό σε συμμόρφωση μάλλον παράλληλα και όπως ισχύει και για τα συστήματα θεωρήσεων. Οπότε έτσι να ε, μπορούμε από τη βάση των αποτυπωμάτων να εντοπίσουμε κάποιον ο οποίος παραμένει και διαμένει παρανόμως και να συνεργαστούμε με τη βάση αυτών των στοιχείων με την χώρα προέλευση επίση και την αναγνώριση προσώπου, να έχουμε το αντίστοιχο λογισμικό και να μπορούμε να κάνουμε ό,τι συγκρίσει χρειάζονται για περιπτώσει που δεν έχουμε ή ποιοτικά ή δεν έχουμε καθόλου αποτυπώματα για να μπορέσουμε να κάνουμε την ε, ταύτιση και να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια να αξιοποιηθεί αυτή η φωτογραφία, αυτή η λήψη της εικόνας του προσώπου. Επίσης για τους ετούντες ε, διεθνή προστασία, είπαμε υπάρχει η ίδια περίοδος αποθήκευση και διακράτησης, δηλαδή 10 χρόνια όπως είχε και τώρα, άρα να ισχύσει η δεκαετία και για αυτές τις καινούργιες κατηγορίες των παρανόμων ε, μεταναστών, αλλά ε, για κάποιες αυτές τις κατηγορίες να έχουμε πέντε αιτία. Με λίγα λόγια αυτά περιέχουν οι προτάσεις μας και ό,τι ερωτήσεις έχετε να σας απαντήσω. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κυρκόπη είναι ο εισηγητής μας για την έκθεση αυτή. Δυστυχώς δεν θα μπορέσει να παραστεί σήμερα. Θα πάρει όμως το λόγο ανταυτού η κυρία Στίβενς, η οποία και παίρνει το λόγο παρά αυτά. Thank you, Chair. Uh, dear Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αντικαθιστώ τον Τίμωθη Κύρκο, ο οποίο ε, δεν ε, μπορεί να προσέλθει στη συνεδρίαση σήμερα. Υποστηρίζουμε πλήρως ε, την πρόταση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής και θεωρούμε ότι όλα τα στοιχεία είναι απαραίτητα σε ό,τι αφορά το σύστημα ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ECR, η ομάδα του ECR θεωρεί ότι η συμπερίληψη των βιομετρικών στοιχείων αποτελεί μια βελτίωση για να πετύχουμε ε, μια μεγαλύτερη ακρίβεια και αποδοτικότητα του συστήματο, αλλά φυσικά θα πρέπει να συνάδουν με τα εφιστάμενα πρότυπα για προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να έχει εμπιστοσύνη στο ίδιο σύστημά τη για το άσυλο και να εξασφαλίζω ότι θα επιστρέφονται οι παράνομα διαμένοντες εδώ, θα πρέπει να έχουμε σύγχρονα και διαλειτουργικά συστήματα και μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Το ECR υποστηρίζει λοιπόν την ανάγκη να επεκταθεί η περίοδος διατηρήσης ε, στο σύστημα, γιατί 18 μήνες πολύ απλά δεν αργούν για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα σε ευρύτερο επίπεδο και για να υπάρχει τα λειτουργικότητα του συστήματος του Eurodact με τα άλλα συστήματα και να βελτιωθεί συνολικά το σύστημα ασύλου της Ένωσης όπως ε, τονίζει και πολύ σωστά η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε, άλλες, σε τομείς ε, η κλασική περίοδος διατήρησης των δεδομένων είναι πέντε χρόνια. Μας φαίνεται σωστό αυτό το διάστημα. Τέλος, το το ζήτημα της συλλογής αποτυπωμάτων, ακτιλικών αποτυπωμάτων των ανηλίκων. Προ το παρόν το όριο αυτό είναι στα 14 χρόνια. Το ECR έχει ζητήσει πιο χαμηλό χρονικό όριο και πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί μεγαλύτερη και επιτελικότερη ανάγκη τώρα. Μπορεί να πέσει λοιπόν από το όριο στα 6 χρόνια από την ηλικία αυτή και μετά με μια κάποια σχετική ακρίβεια μπορεί να γίνει αναγνώριση του παιδιού. Το πιο σημαντικό όμως στοιχείο είναι όπου, ότι έχουμε μια κατάσταση με εκατοντάδες χιλιάδες ε, μη ταυτοποιημένους ανηλίκους ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδεχομένω από ό,τι μας λένε οι ειδικοί να αποτελεί η συλλογή Δεκφυλικών Αποκτημάτων μια λύση για την καλύτερη προστασία του, ιδιαίτερα σε περίπτωση αγνοούμενων παιδιών. Και φυσικά αυτό θα πρέπει να γίνει με πάσα ευαισθησία και προστασία προσωπικών δεδομένων. Αν ωστόσο μακροπρόθεσμα αυτό καταφέρει να προστατεύσει τα παιδιά από του διακινητέ, από την εκμετάλλευση, σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Στίβεν, λέει ο Πρόεδρο. Ο κύριος Λέωνας είναι ο εισηγητής από το ΕΛΚΑ. Πάρτε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, θα είναι και σύντομο. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση και συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπε η συνάδελφος από το ECR και θεωρώ ότι αποτελεί αυτή η πρόταση μια σημαντική βελτίωση σε ό,τι αφορά το αναθεώρηση της οδηγίας για τη Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά επικόστρα των χωρών που δεν έχουν ζητήσει διεθνή προστασία και σε ό,τι αφορά τη μείωση του χρονικού ορίου σε 6 χρόνια, στα έξι χρόνια. Και έγινε και μια κράση πριν από δύο εβδομάδες για τους αγνοούμενους ε, ανηλίκους. 20.000 παιδιά αγνοούνται. Είναι λοιπόν ε, επιτακτική ανάγκη να μπορούμε να τα ανοιχνεύουμε καλύτερα. Έχουμε και την Europol, έχουμε και τις ΜΚΟ, μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που συμφωνούν. Ας την εκμεταλλευτούμε για να ρίξουμε αυτό το όριο ηλικία. Σε ό,τι αφορά την περίοδο τώρα διατήρηση των στοιχείων αυτών, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε κάποια καλά βήματα προ τα εμπρό. Να συζητήσουμε βέβαια και την χρονική διάρκεια, αλλά θα βρούμε συμφωνία. Χαίρομαι επίση ε, με την ιδέα να προσθεθεί συστήματα αυτοποίηση ε, προσώπου, πέρα από την ταυτοποίηση μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων. Ερωτώ όμως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι ελάχιστες προδιαγραφές θα προτείνετε σε ό,τι αφορά την αναγνώριση εικόνας αυτή. Θα είναι της διάστατη, την οποία αυτή που γνωρίζουμε δηλαδή ω σήμερα. γνωρίζοντα γνωρίζοντας φυσικά ότι δεν λειτουργεί πάντα καλά. Έχει δυνατότητα επιτυχία και αναγνώριση 50-60% ή θα προταθεί κάποια πιο η οποία θα προταθει καποια πιο συγχρονη τεχνολογια τρισδιαστατη ενδεχομενω η οποια θα αποτελεσει και μία λύση μακροπρόθεσμα στο μέλλον. Πείτε μας λοιπόν δύο λόγια για τον ορισμό του λογισμικού και του υλικού για την ταυτοποίηση προσώπου και εικόνας. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά είναι τα πρωτοκρατικά με σχόλια. Ευχαριστώ κύριε Λένος. Άλλοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Η Προεδρία των Καταφορών. Αν όχι, κύριε Νίλσεν, καλείτε σύντομα να απαντήσετε στους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω απάντηση στην ερώτηση αυτή. Γιατί θα πρέπει η Λίζα να αναπτύξει τη σχετική μελέτη, όχι μόνο για την ανάπτυξη του λογισμικού, αλλά και την κατεύθυνση που θα πρέπει να επιδιώξουμε. Δεν είμαστε λοιπόν ακόμη σε επίπεδο, έχουμε ξεκινήσει και να έχουμε αρκετές πρώτες απαντήσεις. Πάντως θα σημειώσω τις ερωτήσεις σας και θα τις διαβιβάσω, ώστε να σας απαντήσουν όταν είναι έτοιμοι. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό θέμα, είναι θέμα προτεραιότητας αγαπητοί συνάδελφοι και καλό τις λοιπές πολιτικές ομάδες να ορίσουν σκιώδεις ηγητές και να ενημερώσουν τη γραμματεία της Επιτροπής μας το ταχύτερο δυνατό για τα ονόματα. Και αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, περνώ στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που έχει να κάνει με, την Ευρωπαϊ... με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Η Επιτροπή παρουσίασε στις 4 Μαΐου ένα πρώτο σύνολο προτάσεων για τη μεταρρύθμιση του ε, κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, ΣΕΑΣ, αναθεώρηση των κανονισμών Δουβλίνου και Eurodac, καθώς και αναθεώρηση του κανονισμού που θεσπίζει το ε, Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, ΕΑΣΟ. Ο κύριος Νίλσεν είναι εδώ παρόν για να παρουσιάσει την πρόταση μεταρρύθμισης του ΕΑΣΟ που θα αναπτύξει πλήρως καθήκοντα Ευρωπαϊκού Οργανισμού και έτσι διευκολύνει την υλοποίηση και βελτιώνει τη λειτουργία του συστήματος του κοινού συστήματος ασύλου, Ο κύριος Νέλσεν θα λάβει το λόγο πρώτος. Συγητής είμαι εγώ, αλλά θα μιλήσω μετά από σας. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Όπως είπατε πολύ σωστά, ε, στόχος είναι ο οργανισμός ΕΑΣΟ να μετατραπεί σε μια πλήρους λειτουργίας υπηρεσία από τον κανονισμό το 2011 δεν έχει γίνει μεταρρύθμιση της νομικής βάσης μέχρι τώρα. Η ΆΣΟ έχει αρχίσει να αναπτύσσεται και ως την πραγματογνωμοσύνη, τη λειτουργία αλλά και την υποστήριξη των κρατών μελών που στηρίζονται σε αυτήν, σε διάφορα ε, λειτουργίες σχετικές με το άσυλο και θα μπορούσαμε να πούμε ότι η υποστήριξη που προσφέρεται πλέον στην από τα κράτη-μέλη ξεπερνά την εντολή της στο στάδιο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη σε πλήρης διαστάσεις ενός ευρωπαϊκού οργανισμού για το άσυλο και έτσι τα κράτη-μέλη και κατά την υλοποίηση του κεκτημένου του ασύλου αλλά και κατά την ανάπτυξη δράσεων σε σχέση με το συνολικό σύστημα ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν την υποστήριξή της ώστε να είναι ομοιόμορφο για όλους. Θα ήθελα να τονίσω κάποια νέα στοιχεία από αυτά που προτείνουμε. Προτείνουμε ο οργανισμός ΕΑΣΟ στο μέλλον να ετοιμάζει τεχνικού χαρακτήρα έγγραφα, όπως σε παραδείγματι λειτουργικές προδιαγραφές, καταφυντηρίες γραμμές για τη λειτουργία του συστήματος γλου που έτσι θα βοηθούν τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου στον τομέα αυτών για την ε, ε, ο πιο ομοιόμορφη εφαρμογή από τα κράτη-μέλη σε επίπεδο εθνικό των ευρωπαϊκών διατάξεων. Θέλουμε να προχωρήσουμε και σχετικό με το προηγούμενο είναι στη σύγκληση με το, την εφαρμογή, ως προς την εφαρμογή του συστήματος εγκρίσεως ε, της Ε, Άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε πιο πολλή δουλειά σε σχέση με τις πληροφορίες σχετικές με τη χώρα προελεύσεως, ε, ε, κατάρτιση εκθέσεων, παροχή πληροφοριών σχετικές με τη, σχετικών με τη χώρα προελεύσεως που θα διατίθεται στα κράτη-μέλη. Επίσης, ο οργανισμός μπορεί να υποστηρίζει και εμάς την Επιτροπή αλλά και τα άλλα θεσμικά όργανα σε σχέση με μελλοντικού ε, κοινού καταλόγους ασφαλούς χώρας προελεύσεως που όπως γνωρίζετε επίσης ε, βρίσκεται σε εκκρεμότητα σε μια απόφαση που θα πέρασε από το Κορεπέρ. Ε, μετά την έκθεση ΑΣΟ, λοιπόν, θα προχωρήσει η ΑΣΟ και στην αξιολόγηση και την εκτίμηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών με το κεκτημένο. Αυτό θα γίνει και με νομοσύνε, με επισκέψεις δηλαδή στις χώρες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες που επικρατούν εκεί, αλλά και με επαλήθευση περιπτώσεων ε, για να εξεταστεί πώς σε μεμονωμένες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη έχουν υλοποιήσει το κεκτημένο, από την οποία βέβαια θα προκύψουν και συστάσεις προς τα κράτη-μέλη για να προσαρμόσουν ε, την εφαρμογή του κεκτημένου και βέβαια ε, εντοπισμό αναγκών βάσει των οποίων θα μπορούσε το ΕΑΣΟ να υποστηρίξει και να προσφέρει τη βοήθειά του στα κράτη-μέλη. Εν τέλει δε, ο ρόλος του ΕΑΣΟ για την παροχή και τεχνικής υποστήριξης προς τα κράτη-μέλη, αυτό που ονομάζουμε ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη της πρώτης γραμμής που έχουν τον πολύ μεγάλο αριθμό, τον μεγαλύτερο αριθμό ετήσεων ασύλου, όπου ήδη δραστηριοποιείται το ΕΑΣΟ στα όρια των δυνατοτήτων του και θα θέλαμε να ενισχύσουμε αυτές τις διατάξεις πρώτα απ' όλα για να διευκρινιστούν οι όροι ε, των όσων μπορούν να όσα μπορεί να πράξει το ΕΑΣΟ, να υπάρχει ένα σαφές λειτουργικό σχέδιο για τις δράσεις του, αλλά και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις των κρατών μελών, ώστε να προσφέρουν τις πληροφορίες που χρειάζεται το ΕΑΣΟ για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του και να ε, στηρίζει τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι μια πολύ στενή επισκόπηση, ωστόσο. Προτείνουμε, όπως είπαμε, την ανάπτυξη του ΑΣΟ σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με στη θέσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ και θα μου επιτρέψετε και εμένα να κάνω κάποιες σύντομες ε, παρατηρήσεις για το θέμα αυτό. Από ό,τι γνωρίζω, η ΑΣΟ θα πρέπει να προχωρήσει ως ε, καταρχήν συντονιστής του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου προκειμένου να εξασφαλίσετε εκείνη εφαρμογή των όρων του συστήματος. Έχουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου που θέλουμε να γίνει πραγματικά ευρωπαϊκό και ως εκ του ο οργανισμός ασύλου θα πρέπει να ε, μετατραπεί από έναν οργανισμό που συνιστά ε, απλώς σημείο συνάντησης πολλών ε, υπαλλήλων και εκπροσώπων των κρατών μελών σε έναν ανεξάρτητο ευρωπαϊκό οργανισμό που θα προσφέρει υπηρεσίες ιδιαίτερα προς τα κράτη που ε, έχουν τα εξωτερικά σύνορα. Άρα χρειάζεται και τους ε, ανθρώπινους αλλά και τους υλικούς σπόρους, βράχη, μέσο και μακροπρόθεσμα, ε, απαραίτητους για να επιτελέσει το έργο του. Από την ίδρυση ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος μετεγκατάστασης και εγκατάστασης σε θελασσιακούσια βάση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει ε, στο διευκολυντικό ρόλο που διαδραματίσει ο οργανισμό ασύλου ώστε να εξασφαλίσει υψηλότερα ποσοστά συμμετοχή στο πρόγραμμα εγκατάσταση και ιδιαίτερα για τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει στην εγκατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο του ΕΑΣΟ για την καλύτερη υλοποίηση τη εξωτερική διάσταση του κοινού συστήματος ασύλου. Ο κανονισμός, η εντολή, ορίζει μια εντολή για την ΕΑΣΟ έτσι ώστε να ε, συλλέγει και να δρομολογεί δεδομένα ε, όσον αφορά τις αφήξεις υπηκόνων τρίτων κρατών που μπορεί να σημάνουν σημαντικές πιέσεις στα συστήματα ασύλου και υποδοχής με μια ταχύ ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπό τη νέα πρόταση η, υπηρεσία του Ευρωπαϊ... η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασύλου θα πρέπει να ε, εξασφαλίζει την υποστήριξη για την υλοποίηση της νομοθεσίας και ιδιαίτερα θεσπίζοντας ε, κλίδες αναφοράς για την κατανομή των ετούντων το άσυλο υπό τον διορθωτικό μηχανισμό κατανομής και προσαρμογή και με προσαρμογή των ε, στοιχείων με βάση την ετήσια ε, κλίδα κατανομής αλλά και τα ετήσια δεδομένα της Eurostat. Καθώς βρίσκεται υπό επανεξέταση το ισχύον σύστημα Δουβλίνου, μία λύση θα ήταν να θεσπιστεί μια, ένα κεντρικό σύστημα συλλογής αιτήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα μπορούσε να αναπτυχθεί υπό την αιγίδα και την, ε, το κύρος του ΕΑΣΟ. Έτσι κάποιος ο οποίος αιτείται άσυλο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύνολο και όχι από ένα μεμονωμένο κράτο μέλο και αναλόγω θα, γίνεται, θα, θα γίνεται η κατανομή των ευθυνών για οποιονδήποτε ετούντο το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλι ε, μόλις ξεκινάει αυτή η δουλειά. Ως εισηγητής όμω θα προσπαθήσω να συνεργαστώ στο δυνατόν πιο στενά με όλου του σκιώδεις εισηγητές. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε όλοι μαζί να παρουσιάσουμε μια πολύ καλή έκθεση. Μια έκθεση η οποία θα κοιτάει προ τα μπρος, θα μα επιτρέψει να προχωρήσουμε με ασφάλεια στο μέλλον. Και ο κύριο Κοέλιο, από ό,τι βλέπω, σκιώδη ηγητή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, θα ήθελε να λάβει το λόγο. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Τα πορτογαλικά θα σα τα πω, Πρόεδρε λέει ο κύριο Κοέλιο. Πρώτα πρώτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πληρέστατη ενημέρωση από τον κύριο Νίλσον. Ευχαριστώ και τον κύριο Νίντερ Μίλλερ για τα καλά του λόγια στην εισήγησή του. Θα υπάρξει πνεύμα συνεργασίας επομένως μεταξύ μας. Έχω δύο σχόλια προσαγωγικά να σας αναφέρω. Πρώτα-πρώτα, ε, βέβαια και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να θεσπίσουμε και να αποκτήσουμε ένα κοινό σύστημα ασύλου. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι πάρα πολλά κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν αναδεχθεί στο εσωτερικό τους δίκαιο το κεκτημένο. Πρέπει επίσης το ισχύον σύστημα να βελτιωθεί. Επίσης θα πρέπει οι διατάξεις ε, εθνικού δικαίου να εναρμονιστούν σε όλα τα κρατη αλλά και οι πρακτικές των κρατών μελών. Να, γιατί χρειάζεται μια τέτοια υπηρεσία και ένα κοινό σύστημα ασύλου. Οπότε η υπηρεσία αυτή θα υποπτεύει την λειτουργία και τον συντονισμό. Χρειάζεται, επομένως, έχουμε διαπιστώσει ένα θεσμικό πλαίσιο πιο στεγανό. Η ΕΑΣΟ, επομένως, θα γίνει η υπηρεσία που θα έχει αναβαθμισμένες αρμοδιότητες και θα έχει στην διάθεσή της μέσα και πόρους περισσότερα. Οπότε θα υπάρξουν έτσι καλύτερες ε, εγγύσεις για λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Οπότε θα είναι καλύτερα τα πράγματα, όποτε αυξάνονται οι πιέσεις στα μέτωπα των αρμοδιοτήτων. Ε, για άλλη μια φορά ευχαριστώ τον Ιντερ Μίλλερ, αλλά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι θα είναι θετικές οι εξελίξεις Πίτερ, πιστεύω ότι θα πάνε τα πράγματα πολύ καλά στη συνεργασία μας. Ευχαριστώ εγώ, κύριε Κοέλιο. Λέει ο πρόεδρος, θέλει κάποιος συνάδελφος το λόγο. Μήπως η Ολλανδική Προεδρία ή ο κύριος Νίλσεν, όχι από ό,τι φαίνεται. Αφού δεν θέλει κανείς το λόγο, τότε προχωρούμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Πρόκειται για τον κατάλογο των χωρών υπήκο των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρηση διαβατηρίου για διέλευση εξωτερικών συνόρων και επίση ε, για του υπηκόστου των χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. Εισηγητής είναι ο κύριο ε, Δίαθ του Λαϊκού Κόμματο. Και επίση κυρία Γιώτοβα και έχουμε τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάργηση κάποιων θεωρήσεων διαβατηρίου, οπότε και προτείνουν την κατάργηση του μηχανισμού αναστολής, όπως ονομάζεται του κανονισμού 539 του 2001, εκεί όπου ε, εν παρατήματι έχουμε τον κατάλογο των ε, χωρών υπήκο των οποίων θα πρέπει για διέλευση του Σέγγεν να έχουν τη θέση διαβατηρίου. Αυτό ο οργανισμός ε, θεσπίστηκε με τον κανονισμό αυτόν του 2013 και υπάρχει επίση και ένα μηχανισμό αμοιβαιότητα αντίστοιχο. Οπότε είπαμε ότι έχουμε τον ε, εισηγητή μα τον κ. Διά Δεμέρα, ο οποίο επίση είχε αναλάβει και την έκθεση για του οργανισμού το 2013. Δυστυχώ όμω, σήμερα δεν μπόρεσε να παραστεί και θα τον αντικαταστήσει ο κύριος Κοέλιο. Κύριε Κοέλιο, θα θέλατε να αρχίσουμε με εσά ή να, να αρχίσουμε την Κομισιόν. Α, ναι, ε, δεν έχει έρθει όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, άρα εσείς αναγκαστικά θα μιλήσετε πρώτος. Ladies and gentlemen, colleagues, the Commission has arrived. Welcome. Uh, Κατέφτασε η Επιτροπή Συνάδελφοι και μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε έτσι την ε, συνεδρίαση. Είμαστε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Κατάλογος τρίτων φορών. <coughs> και όπως σας είπα, ο κύριος Δίας Δαμέρα είναι ο εισηγητής ε, ναι. για το θέμα αυτό. Ήταν και εισηγητής το 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού. Δυστυχώ όμως δεν θα μπορέσει να παραστεί σήμερα. Θα τον αντικαταστήσει ο κύριος Κοέλιο. Κύριε Κοέλιο, πάρτε το λόγο αν θέλετε και στη συνέχεια θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους συναδέλφους όπως είπατε, μιλάω εξ ονόματος του συναδέλφου Διαστεμέρα, ο οποίος και είναι ο εισηγητής για το θέμα αυτό, δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα στη συνεδρίασή μας. Έχει υποχρεώσει στην Ισπανία, ζητά συγγνώμη για το γεγονός αυτό. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τον εισηγητή, το θέμα αυτό θα αποτελέσει προτεραιότητα. Θα εργαστούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται τη σημασία του μηχανισμού αναστολής για την πολιτική για τις θεωρήσεις. Ο κ. Διεθμέρα. θα παρακολουθήσετε την έκθεση αυτή και θα ακολουθήσει το εξή χρονοδιάγραμμα. Σήμερα έχουμε την παρουσίαση λοιπόν στην Ευρωπαϊκή. Προγραμματίζεται συνάντηση των σκιωδών για την 31η Μαΐου και η παρουσίαση θα γίνει η παρουσίαση του προγράμματος εργασίας. 15 Ιουνίου παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης. 30 Ιουνίου παρουσίαση στη λίβε Και κατά πάσα πιθανότητα 12 Ιουλίου θα έχουμε ψηφοφορία στην Επιτροπή μας, στη ΛΥΜΠΕ. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα, αυτό είναι το πρόγραμμα που προτείνει ο Είσαι Δία Δομέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοέλιο, και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο πρώτα-πρώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μα παρουσιάσει την πρόταση. Μετά θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψει. Η κυρία Γκαγέγο Καλσίλτα έχει το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και καλησπέρα. Θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση τη πρόταση που ανέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4 Μαΐου για την αναθεώρηση του μηχανισμού αναστολής. με την αναθεώρηση του 2013 με τον ε, κανονισμό 129. Δεδομένη τη κατάσταση τη μεταναστευτική ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και την ολοκλήρωση κάποιων διαλόγων και πραγματεύσεων για την απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων όπως η Γεωργία, Κοσμοπέδιο και Τουρκία. Δεδομένων λοιπόν όλων αυτών, κάποια κρατημέλη αναρωτιούνται κατά πόσο το σύστημα το οποίο προβλέπεται δίνει την απαραίτητη ευελιξία για ταχύτατη αντίδραση σε κατεπίκουσες περιπτώσεις σε ό,τι αφορά αναστολή της εξαίρεσης της υποχρέωσης για τις θεωρήσεις κάποια από τα θέματα τα οποία εντοπίστηκαν ως ε, βασικά ενδεχόμενα ελαττώματα του εφιστάμενου μηχανισμού και μπορείτε να δείτε πιο πολλές πληροφορίες στο σχετικό μνημόνιο, είναι τα εξής. Καταρχάς, είναι περιορισμένες ε, οι περιπτώσεις όπου μπορεί να γίνει τέτοια αναστολή. Δεν περιλαμβάνεται η έλλειψη συνεργασία, ε, για παράδειγμα, από πλευρά τη τρίτη χώρα για την επανειστοχή των επικών τη χώρα αυτή. Και όπω ξέρετε, σε άλλε περιπτώσει προβλέπεται, μάλλον προβλέπεται η αναστολή λόγω έλλειψη συνεργασία ε, σε ό,τι αφορά του δικού μα επικού, όχι όμω αυτών των τρίτων χωρών. Κάτι άλλο. Ότι ο μηχανισμό αυτό μπορεί να ταθεί σε εφαρμογή μόνο από τα κρατημέλη, κάποια κρατημέλη προτείνουν να μπορεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τον κινητοποιήσει τον μηχανισμό αυτό. Ένα τρίτο ζήτημα το οποίο αναφέρθηκε είναι η περίπτωση αναφοράς και οι πρόθεσμίε για την εφαρμογή του υφιστάμενου μηχανισμού ήταν υπερβολικά μεγάλες και έτσι δεν μπορεί να υπάρχει μια γρήγορα αντίδραση σε καταπήγουσα ανάγκη μετά από τις συζητήσεις διαπραγματεύσεις ε, με τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παρουσιάσει μια τροποποίηση του 539 και σε ό,τι αφορά ίδρα το Κωσυφοπέδιο και την Τουρκία. Και βασικός λοιπόν στόχος της πρότασης είναι να ενισχυθεί ο μηχανισμός αναστολής, να είναι πιο εύκολο για τα κράτη-μέλη να ορίσουν τους όρους και τις περιπτώσεις που θα οδηγήσουν σε αναστολή και να μπορεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινητοποιήσει τον μηχανισμό. Σε ό,τι αφορά την, η, τη μείωση της περίοδου προθεσμίας αυτής της περίοδου που προβλέπεται, όπως ξέρετε, η πρόταση ε, μάλλον η περίοδος αυτή ανέρχεται σε έξι μήνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να μειωθεί σε δύο μήνες. Μετά την ε, κοινοποίηση από τα κρατημέλη, η, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τρεις μήνες στη διάθεσή της ε, για να ε, προβεί σε πράξη έγκρισης. Τώρα προτείνεται αυτή η τριμηνία περίοδος, η τριμηνή περίοδος να γίνει περίοδος ενός μήνα. Μία άλλη περίπτωση κοινοποίηση επίση προτείνεται σε ό,τι αφορά τον αριθμό απορριφθέντων προτάσεων επανεισδοχής. Άρα όχι μόνο έλλειψη συνεργασίας του τέτοιου κράτους, της τρίτης χώρας, αλλά και έλλειψη ε, συνεργασίας ό,τι αφορά τη τρίτη χώρα και σε ό,τι αφορά του ε, τους ε, τη της χώρας που έχουν μπει. Τέλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν λάβει συγκεκριμένα στοιχεία για α, τέτοιες περιπτώσεις ή αν κάποια χώρα δεν συνεργάζεται σε θέματα επανεισδοχής, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της τρίτη χώρα. Υπάρχουν και άλλες ε, πιο μικρές αλλαγές σε ό,τι αφορά την σε 7 χρόνια της περίοδου κατάργησης και αυτές είναι ουσιαστικά οι αλλαγές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζουμε δε και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να συμφωνήσουν και να δοθεί ασφαλώς προτεραιότητα στο θέμα αυτό για να εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν και να παρουσιαστεί παράλληλα με το θέμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Η συζήτηση δε για το θέμα αυτό δεν θα πρέπει να καθυστερήσει τις συζητήσεις τις άλλε. Γι' αυτό χαιρόμαστε που έχει μπει ήδη στην ημερησία διάταξη το θέμα για το κοσμοπέδιο και τις άλλες χώρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα λοιπόν να ρωτήσω κατά πόσο θέλει κανένα συνάδελφο να πάρει το λόγο. Η κυρία Στήμενς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και συνάδελφοι. Η αντιπροσωπεία μου του NVA πιστεύει ότι χρειαζόμαστε έναν πιο ισχυρό μηχανισμό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, συμφωνίες για την απελευθέρωση των θεωρήσεων που αποτυγχάνουν. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία δεν υπήρχε πλειοψηφία. Αυτό ε, όμως πλέον έχει επιτευχθεί και την πρόταση αυτή λοιπόν την εισάκουσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι ενισχύει το σχετικός μηχανισμός με κάποιο βαθμό αυτοματοποίησης, πιο σύντομες χρονικές περιόδους και πιο αυστηρούς όρους, καταφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει ε, πιο πολλές δυνατότητες κινητοποίησης του μηχανισμού. Σε περίπτωση που δεν γίνεται αποδεκτή συμφωνία για την επανεισδοχή υπηκών των χωρών, οπότε υπάρχει θέμα ασφάλεια και σε περιπτώσεις που οι χώρες που έχουν λάβει την εξαίρεση ε, δεν σέβονται πλέον ε, τα benchmarks που θα δικαιολογούσαν τη διατήρηση τη εξαίρεση. Αυτό που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εξή. Ε, ακούσαμε και τι έχει γίνει με την κυβέρνηση Τουργάν. Θα πρέπει να μπορούμε από ευρωπαϊκή άποψη να επιδείξουμε και την ισχύ μα και να θέσουμε του όρου μα. Και δεν θα πρέπει να αφαιθούμε τελείω και να αφήσουμε την τύχη μα τελείω στα χέρια του Ερντογάν. Θα πρέπει όλα, αν χρειαστεί, να θέσουμε όλα τα θέματα και άλλε περιπτώσει απελευθέρωση θεωρήσεων σε αναμονή. Πέρα από τους ε, από τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρεί το Κωσοφοπέδι, η Ουκρανία και οι άλλες χώρες σήμερα. Thank you very much, uh, Ευχαριστώ, κυρία Στίβενς. Άλλα σχόλια, παρακαλώ. Παρατηρήσεις. Τότε παρακαλώ την κυρία Καγιέκου. Αν θέλει να απαντήσει, όχι. Πάλι εύκολο θέμα. Και πάμε στο επόμενο. Κατάλογος τρίτων χωρών, η υπήκοη των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση θεωρήση για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και κατάλογος τρίτων χωρών, η υπήκοη των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. Κουσφοπέδιο. Η κυρία Φαϊόν είναι η συγγήτρια και θέλω απλώ να υπενθυμίσω, συνάδελφοι, ότι το πρώτο θέμα έχει να κάνει με την μεταφορά του κοσμοπεδίου στον κατάλογο των χωρών για τις οποίες δεν απαιτείται θεώρηση διαβατηρίου, δηλαδή τις χώρες ε, στην κατηγορία του βιομετρικού διαβατηρίου. Πρόκειται για μια μακρά διαδικασία που ξεκίνησε υπό τη διαδικασία του διαλόγου για την απελευθέρωση από τη θεώρηση ε, τον Ιανουάριο του 2012 μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κωσυφοπεδίου. Ο διάλογο αυτό ε, διεξήχθη χωρί, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των θέσεων των κρατών μελών στο καθεστώ και την αναγνώριση του Κωσυφοπεδίου. Από την εκκίνηση του διαλόγου για τη θεώρηση των διαβατηρίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή μα για την τήρηση από πλευρά του Κωσυφοπεδίου και την εκπλήρωση των προποθέσεων για την απελευθέρωση τη θεώρηση. Στην τέταρτη και τελευταία έκθεση προόδου που υιοθετήθηκε στις 4 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εξέφρασε τη θέση ότι το, κοινοβου... ότι το κοσμοσυφοπαίδιο έχει εκπληρώσει τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις με βάση και τη συνεννόηση ότι την ημέρα της υιοθέτησης αυτής της πρότασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το κοσμοσυφοπαίδιο θα έχει κυρώσει τη Συμφωνία Συνόρων με το Μαυροβούνιο και θα έχει ενισχύσει την καταγραφή ε, και τις επιδόσεις ως προς την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Ε, με βάση αυτή την αξιολόγηση, λοιπόν, η Επιτροπή προτείνει την ε, πρόταση που έχετε ενώπιόν σας με την τακτική νομοθετική διαδικασία. Η κυρία Φαγιόν απουσιάζει δυστυχώ, είναι η εισηγήτρια. Θα την αντικαταστήσει η κυρία Λαουριστίν, στην οποία δίνω τον λόγο πρώτα και μετά θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Η Τάνια με παρακάλεσε να σας παρουσιάσω τη δήλωσή της, την Αναγιγνώσκο λοιπόν, εξ ονόματος της Τάνια, η οποία λέει «Αγαπητοί συνάδελφοι, Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστώ την Επιτροπή για την παρουσίαση μιας ε, αναμενόμενης από καιρό και ευπρόσδεκτης πρότασης. Έχω την ε, ευτυχία να συνεχίσω ένα επιτυχές ταξίδι που ξεκίνησαν πριν από 5-6 χρόνια άλλα δυτικά, κράτη των Δυτικών βαλτοκανίων και έτσι το Κωσυφοπαίδιο ε, το οποίο ήταν απομονωμένο λόγω του καθεστώτος θεώρησης των διαβατηρίων, είχε μείνει μόνο του. Πρόκειται για μια έκθεση και μεταρρύθμιση η οποία απαιτείται, πρέπει να προχωρήσει γρήγορα ώστε να μην χάσει κάθε ελπίδα για μελλοντική συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο κοσφοπέδιο. Αποτελεί εγγύηση σταθερότητας και κινητήρια δύναμη για μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται ε, στη χώρα. Επίσης είναι πολύ σημαντική η απόφαση για την απελευθέρωση από την υποχρέωση θέωση του διαβατηρίου για τους πολίτες γιατί αποτελεί ένα από τα σαφέστερα επιτεύγματα μιας χώρας εν ώψη του μέλλοντος. Δεν πρέπει να σταματήσουμε λοιπόν την προσπάθεια, πρέπει να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες και τις ελπίδες των πολιτών. Ε, αυτό θα διευκολύνει όχι μόνο τις διαπροσωπικές επαφές αλλά και εκπαιδευτικέ ανταλλαγές, πολιτισμικές και άλλες. Ταυτόχρονα όμως θα βγάλει εκτός δικτύου και παιδείας όποιον εγκληματία έχει εκμεταλλευτεί την κατάσταση που ισχύει τώρα. Και νομίζω ότι το κοσμοπέδιο θα ε, ε, επιστεγάσει με επιτυχία αυτή του την προσπάθεια. Πιστεύω ότι θα είναι σύντομα δυνατό και για του πολίτες του να υποφεληθούν από όλα τα ωφέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσβλέπω σε καλή συνεργασία με του συναδέλφου από το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο, αλλά και του φίλου από το Κοσμοπεδίο. Μέχρι τώρα είχαμε πολύ καλή συνεργασία και σχέσει με ε, όλου του εμπλεκόμενου. και πιστεύω ότι αυτό θα συνεχιστεί. Στόχος είναι να εγκαθιδρυθεί μια, ένα θεματολόγιο φιλόδοξο για να αντιμετωπιστούν τα εναπομείναντα ζητήματα και παρακαλώ αντίστοιχα να κάνει το ίδιο και το Συμβούλιο. Εν τέλει, έχω ένα σχόλιο μόνο ή μάλλον τροφή για σκέψη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνω θα ήθελα σε ευρύτερη προοπτική και υπό εξέταση να τεθεί το ζήτημα των επιμέρους προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρεί κάθε χώρα για να της χορηγηθεί η απαλλαγή από τη θεώρηση του διαβατηρίου. Ορισμένες έχουν τεχνικό χαρακτήρα, κάποιες άλλες όμως προϋποθέσεις είναι πολιτικές και άλλες δεν είναι καν καθαρές, ξεκάθαρες ή και συναφείς με την ισχύουσα πρακτική. Έχουν διευκρινιστεί αρκετές από τις προϋποθέσεις ε, που απαιτούνται, αλλά δεν έχει οριστεί ο τρόπος με τον οποίο αξιολογούνται αυτές. Πώς λοιπόν ορίζει κριτήρια για τρίτες χώρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς αυτά αξιολογούνται. Πώς μπορεί η χώρα όπως το Κοσμοπέδιο να έχει προϋποθέσεις οι οποίες δεν απαιτήθηκαν από το Μαυροβούνιο ή άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στη διαδικασία διαλόγου για την απελευθέρωση από τη θεώρηση του διαβατηρίου. Ε, επ' αυτή την έννοια λοιπόν θα κάνω ό,τι μπορώ για να, ανοίξω, να, να εξετάσω, ανοίξω την εξέταση όλων των εκκρεμών ζητημάτων και να βρεθεί μια λύση αποδεκτή για όλους τους εμπλεκόμενους. Επιστρέφω μόλις από το κοσμοπέδιο μου, εκεί πριν από μία εβδομάδα, ύστερα από μία πρώτη ιστορική ε, συνάντηση ε, και πιστεύω ότι θα μπορέσω όταν τους επισκεφθώ και πάλι να έχω πιο καλά νέα να τους παρουσιάσω για να ενισχυθούν και οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοσμοπεδίου που ε, ακόμα δεν έχουν προχωρήσει ύστερα από την Συμφωνία Συνεργασίας και Εταιρικής Σχέσης. Το Κοσμοπεδίο ανήκει στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, εδώ είναι η θέση του και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Πρέπει να καταστήσουμε το μέλλον πιο λαμπρό και να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί τις μεγάλες προκλήσεις των καιρών μας. Αυτό το οφείλουμε όχι μόνο στους εαυτούς μας αλλά και στους πολίτες του Κοσμοπεδίου και αυτά ήταν τα λόγια της Τάνιας, όχι τα δικά μου. Πέρι το λόγο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κυρία Γκαγέγο Κασίλτα. Ευχαριστούμε και την κυρία στην διότι μας ε, ε, διαβίβασε η συγκεντρία διακίνηση το, ε, την πρότασή είπαμε και στην πρωτοβουλία του 2012 και με αυτό το χαρτί πορεία, με τι προποθέσει που θα πρέπει να πληρούνται, ούτω ώστε να γίνει αυτή η καταργήση θεωρήσεων, οπότε να. Και έχουμε και το θέμα που στο τέλο τη ανακοίνωση του κειμένου, ότι για κάθε χώρα ε, έχουμε χωριστή ε, πρόβλεψη των προϋποθέσεων. Το ίδιο έγινε και με το πεδίο. Άργησε λίγο περισσότερο από άλλε χώρε. Δεν είναι θέμα επομένω ε, συνέπεια εσωτερική πολιτική, είναι ε, το τι γίνεται με κάθε χώρα, τι γίνεται με το οργανωμένο έγκλημα, τι ασφάλεια υπάρχει περί τα έγγραφα κλπ. Υπάρχουν και κάποια κοινά κριτήρια βέβαια, αλλά περιπτωσιολογικά γίνεται ο καθορισμό τη πορεία του κάθε κράτου. Και είπαμε ότι όλα αυτά γίνονται με την επιφύλαξη τη τοποθέτηση ε, των κρατών μελών για το καθεστώς της χώρας και είπαμε ότι έχουμε την αποστολή για το κράτος δικαίου στη χώρα και οπότε ήταν πολύ σημαντικός ο ρόλος της αποστολής του ώστε να βοηθηθεί η χώρα να κάνει κάποιες μεταρρυθμίσεις και έτσι να πληρεί τις προϋποθέσεις που τάση ο της πορεία. Έχουμε τρει εκθέσει την τελευταία τριετία σχετικώ. Φεβρουάριο του 2013, τον Ιούλιο του 2014, αλλά και τον Δεκέμβριο του 2015. Και η τέταρτη έκθεση, όπως είπε ο πρόεδρο, στις 4 Μαΐου μαζί με την πρόταση αναθεώρησης του σχετικού κανονισμού σε αυτές τις τέσσερις εκθέσεις είπαμε ότι το κοσμοπέδιο κάνει σημαντικά βήματα ούτως ώστε να πληρεί ε, τις δύο βασικές προϋποθέσεις που η πρώτη είναι η κύρωση της συμφωνίας με το Μαυροβούνι και τα σύνορα και επίσης η άλλη προϋπόθεση είναι το ότι θα πρέπει να γίνουν βήματα πρόοδος και τα πολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, οπότε επί τη βάση της αξιολόγησής μας με την έκθεση ε, αποφασίσαμε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του χάρτη πορεία διατάρχης θεώρησης. Και βέβαια επί τη βάση του ότι τη μέρα θέσεως σε ισχύ ε, αυτού του νομοθετήματος το κοσμοπέδιο θα έχει κυρώσει αυτή την ε, συμφωνία για τα μεθοριακά με το Μαυροβούνιο και επίση θα έχει αναβαθμίσει ε, το θέμα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος τη σχετική πολιτική. Έχουμε τώρα, είπαμε, την αναθεώρηση του κανονισμού 539-2001, ε, ότι υπάρχει η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτως ώστε από το δεύτερο παράδειγμα, τμήμα 4 του κανονισμού 539 του 2001, συγγνώμη, λέει η από το πρώτο παράδειγμα πάει στο δεύτερο τέλο πάντων, το κοσυφοπαίδιο και καταληκτική παρατήρηση είναι η εξή. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, η τροποποίηση καλύπτει μόνο αυτού που έχουν βιομετρικά διαβατήρια. η ΚΑΟ και τα άλλα διεθνή ε, πρότυπα για την ασφάλεια. Βέβαια χρειάζεται και αμοιβιότητα, αλλά το Κοσμοπέδιο ήδη έχει τηρήσει αυτή την προπόθεση τη αμοιβιότητα για του πολίτε. Ένωση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμεί ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρο. Κυρία Σκρίπικ, εκ μέρου τη κυρία Μακοβέη για την ECR, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Δυστυχώ η κυρία Μακοβέη δεν μπόρεσε να παραστεί σήμερα και ζητάει να την συμπαθούμε για αυτή την αλλαγή τελευταία στιγμή, οπότε θέλει και να σας διαβάσω ποια είναι η άποψή της. Είναι η δική της άποψη, όχι η δική μου. Να σας διαβάσω το μήνυμά της επομένως. Η κατάργηση τις βίζες θα πρέπει να δοθεί μόνο όταν μια χώρα πληρεί απολύτω κάποιες προϋποθέσεις και κάποια κριτήρια τα οποία ορίζονται στο χαρτί πορεία. Στην περίπτωση του Κοσμοπεδίου επιβεβαιώνει η Επιτροπή ότι όντως πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις για ε, την κατάρξη της θεώρηση όπως ορίζονται και στον ε, χαρτί πορεία. Όλα αυτά τα οποία έγιναν από τότε που ξεκίνησε την πορεία του και τη διαδρομή του, διάλογο με τη χώρα για την θεώρηση. πάντω. έχουμε άλλε δύο πάγιε βασικέ προποθέσει που θα πρέπει να πληρώνται πριν καταργηθούν οι θεωρήσει για του υπηκόου τη χώρα. Δηλαδή, η κύρωση τη συμφωνία για την μεθόριο με το Μαυροβούνιο και επίσης θα πρέπει να αναβαθμίσει την αντιμετώπιση του Κόσοβο του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. επίση. επίσης, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει την ε, εποπτεία βάσει του χάρτη πορείας για την ε, συνέχεια και μετά την κατάσταση θεώρησης για αυτούς τους τέσσερις άξονας όσον αφορά την επανένταξη και την επανεισδοχή. Ε, ευχαριστούμε τον πρόεδρο και την κυρία Γκάμπριελ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχόλια που έκανε και για την δήλωση που έκανε και θα πρέπει να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένη που η, η η κυρία Φαγιόν, προτίθεται να συνεργαστεί με την Επιτροπή και με όλους τους συναδέλφους. Δεν έχω δε αμφιβολία ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσπιστούμε όπως πάντα την θέση μας όπως πάντα, λοιπόν, όταν μιλάμε για θεωρήσεις θα πρέπει να μιλάμε και για τον πολίτη. Χρειαζόμαστε πολιτικό διάλογο, χρειαζόμαστε και ένα σαφές μήνυμα προς τους πολίτες του Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο κατά την ανάλυση των τεκτενωμένων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκ παραλλήλου να απευθύνω έκκληση και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε εγκαίρως να λαμβάνουμε τα στοιχεία και τις πληροφορίες. Μόνο αν είναι καλή η συνεργασία μας, θα μπορέσει αυτή η εργασία να σταθεί με επιτυχία σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση από το καθεστώς των θεωρήσεων. Αναφέρθηκε ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια του οδικού χάρτη. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω τέσσερις ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, Πείτε μας, το κοσφοπέτιο έχει δεύτερο δευτερογενή νομοθεσία σε ό,τι αφορά την αλλαγή των ονομάτων. Είναι σημαντικό το γεγονός αυτό για να μην υπάρχουν καταχρήσεις και να μην κυκλοφορούν βιομετρικά διαβατηρία με ανακριβή αναλυθή ονόματα. Αυτό αποτελεί και ένα από τα κριτήρια. Κατά δεύτερον, ο δεύτερος θεματικός ε, τομέας έχει τίτλο «Ενσωματωμένη διαχείριση συνόρων». Ενοποιημένη διαχείριση συνόρων. Έχει αναλύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόγο για τον οποίο είναι χαμηλός ο αριθμός των ε, ασύλων που χορηγούνται σε πολίτες του Κωσυφοπεδίου παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει πολλές αντίσεις και Τρίτον, τι γίνεται με το οργανωμένο έγκλημα. Και τέταρτον, έχω να κάνω μια ερώτηση σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ξέρουμε ότι ο θεσμός του διαμεσολαβητή είναι σημαντικότατος προκειμένου να υπάρχει η εξασφάλιση των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και μία από τις συστάσεις άλλωστε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Κωσυφοπαίδιο ήταν να αναπτύξει τον θεσμό του διαμεσολαβητή τι έχει επιτευχθεί εδώ. Αυτά είναι, αυτές είναι οι πρώτες ερωτήσεις μου βάσει και της έκθεσης που έχουμε λάβει μέχρι τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πραγματικά είναι σημαντικά για μας και θα ήθελα να επαναλάβω και να υπογραμμίσω ότι θέλουμε να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλουμε να λάβουμε πιο πολλά στοιχεία από την Επιτροπή προκειμένου να καταλήξουμε και σε μια οριστική απόφαση βάσει μια σωστή μεθοδολογία η οποία θα αποστείλει και ένα σωστό μήνυμα προ του πολίτε τη χώρα αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε, κυρία Γκάμπριελ. Η Προεδρία, μήπω θέλει να πάρει το λόγο. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστούμε και αγαπητοί ευρωβουλευτές για την πρόσκληση. Το θέμα αυτό θα έχει μεγάλη σημασία και για το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά την τροποποίηση του μηχανισμού αναστολή την προηγούμενη Παρασκευή. Ενέκρινε μια τοποθέτηση για την πρόταση αυτή και το Συμβούλιο ε, είδε και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οποία και σας ευχαριστούμε. Προσέθεσε κάποια στοιχεία σε αυτό σε ό,τι αφορά ένα μηχανισμό παρακολούθησης, monitoring, όπου ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει τη ΣΥΟΣΑ έκθεση προς το Συμβούλιο και την ε, Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την παρακολουθήση των κριτηρίων τα οποία θα πρέπει να βλούν οι χώρε οι οποίες έχουν εξαιρεσει από τις θεωρήσεις και υπάρχουν, έχουν προσθεθεί δύο λόγοι για κινητοποίηση του μηχανισμού αναστολή σε ό,τι αφορά την δημόσια τάξη και την ιστορική ασφάλεια και σε ό,τι αφορά το δικαίωμα επιστροφή και τα άτομα που επιστρέφουν. Και επίσης υπάρχει κάποιο μεγαλύτερο ε, αυτοματισμό για την εισαγωγή αυτή τη περίοδο αναστολή 6 μηνών. Τα κράτη-μέλη τώρα είναι ικανοποιημένα με την ε, συμφωνία που έχει επιτευχθεί και ελπίζουμε σύντομα να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα περιεχόμενα της ε, συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ξεκινήσουμε και διαπραγματεύσεις και προσβλέπουμε και στην ε, τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του μηχανισμού, σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς τώρα για την απελευθέρωση του Κωσυφοπεδίου και της Ουκρανίας συζητήθηκε ήδη μία φορά Δεύτερη φορά προγραμματίζεται συνάντηση και συνομιλία των κρατών μελών με το θέμα αυτό στις 14 Ιουνίου. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρος. Κύριε Αγκαγέγκο Καστίλτα, μήπως θέλετε να πάρετε το λόγο για να απαντήσετε τις ερωτήσεις που έθεσαν τα μέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, για το monitoring, την παρακολούθηση, βεβαίως θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την γύρωση ε, της ε, συμφωνίας ε, για το συνδρόμο με το Μαυροβούνιο και βέβαια της προόδου σε σχέση με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς στο πλαίσιο του μηχανισμού παρακολούθησης μετά την απελευθέρωση όπως ισχύει άλλωστε και για τις χώρες της, ε, για όλες τις χώρες Δυτικών Βαλκανίων. Και ούτως ή άλλως είμαστε σε διαρκή επαφή με τον σύνδεσμό μας με το Κωσοφοπέδιο για τα θέματα αυτά και τα παρακολουθούμε ανεξαρτήτως για την κυρία Γκάμπριελ σε σχέση με, τον, με την νομοθεσία. Για την αλλαγή των ονομάτων έχουμε τη σχετική νομοθεσία την έχουμε υιοθετήσει για τα αιτήματα ασύλου οι παράτυποι μετανάστες, ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών και ετοιμάτων ασύλου έχει από το 2008 μειωθεί ως προς τους υπηκόους του έχει φτάσει σε χαμηλότερα επίπεδα από την κίνηση του διαλόγου την ε, Θεός Νεβατήριο το 2012. Άρα νομίζω ότι αυτή είναι η απάντηση για το διαμεσολαβητή Ε, μπλοκ 4 θεμελιώδη δικαιώματα συγκεκριμένα από τις προϋποθέσεις έχουμε όντως ε, βεβαιωθεί ότι έχει δημοσιονομική ανεξαρτησία ο θεσμός του διαμεσολαβητή και για φέτος έχει στη θέση του έχει προϋπολογισμό 400.000 ευρώ άρα είναι σύμφωνο με τις δεσμεύσεις με το διαμεσολαβητή του οικοσφοπεδίου και πιστεύουμε ότι έτσι θα μπορέσει να επιτελέσει το νέο του έργο με βάσει τα θέματα που είναι στο πακέτο μέτρων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτές είναι κάποιες από τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Άλλες ερωτήσεις ή αντιδράσεις στις δηλώσεις αυτές, αν όχι, τότε θα σας πω μόνο ότι η παρουσίαση του σχεδίου εκθέσεως για το θέμα αυτό προβλέπεται στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ στις 15-16 Ιουνίου και προχωρώ στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι ο κατάλογος τρίτων χωρών υπήκοε των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και τρίτων χωρών υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποκρέωση αυτή η Ουκρανία συγκεκριμένα. 2008 έχει ξεκινήσει ο διάλογο. Από τον Εύρωο του 2010 ένα σχέδιο δράση για την απελευθέρωση τη θεωρία βατηρίων έχει ε, ξεκινήσει και συνεχίζεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει ε, παγίω εκθέσει προοδού στην Επιτροπή μα νύψε μια συμφωνία ε, διευκόλυνσης θεωρήσεων και επανεισδοχής με την Ουκρανία. Ήταν η προϋπόθεση για την κίνηση και τη συνέχιση του διαλόγου για την απελευθέρωση θεώρησης με την Ουκρανία. Στην έκτη και τελευταία έκθεση προόδου που υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει πως η, η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει την απαιτούμενη πρόοδο και έχει υποβάλει την ε, φυστάμενη πρόταση που θα συζητηθεί υπό την τρέχουσα νομική ε, νομοθετική διαδικασία αρμόδια είναι η κυρία Γκάμπριελ ως εισηγήτρια. Της δίνω πρώτη στο λόγο και μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους λοιπούς ομιλητές. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινώντας θέλω να ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία απευθύνεται κατά κύριο λόγο σήμερα η παρέμβασή μου. Καταγράφει λοιπόν ε, τις ε, προόδους στη διαδικασία ε, του διαλόγου για την απελευθέρωση της θεώρησης η Επιτροπή και εγώ θέλω να σημειώσω ότι αυτές οι προόδοι σηματοδοτούν πάνω από όλο για μας τη σημασία της στηρίσης ε, εκ των προτέρων οριστέντων κριτηρίων για το συμφέρον των ίδιων των πολιτών, για την επιβολή κράτου δικαίου, κράτου δικαιοσύνη, ασφάλεια και που εν τέλει οδηγήσουν, πρέπει να οδηγήσουν στην απελευθέρωση από τη θεώρηση διαβατηρίου. Και αυτό δείχνει και την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ουκρανία. Με την παρουσία λοιπόν τη Επιτροπή και πριν από την παρουσίασή τη, θα ήθελα να διατυπώσω κάποιε ερωτήσει, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, οι οποία στη συνέχεια με τι απαντήσει που θα λάβω θα μου επιτρέψουν να προχωρήσω και στη σύνταξη τη εκθέσεω. Μια πρώτη ερώτηση δεδομένη της ε, πρότασης τώρα για την εξαίρεση για τους φέροντες ε, βιομετρικά διαβατήρια. Θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή πόσα τέτοια έχουν εκδοθεί από τι αρχέ τη Ουκρανία. Επίσης, ω προ την ασφάλεια των ε, εγγράφων ταυτοποίηση, υπάρχει μια έκθεση για την αυτοματοποίηση του συνδέσμου μεταξύ του Εθνικού Μητρώου Ληξιαρχείου και του Μητρώου Πολιτών. Ερωτώ λοιπόν πολύ απλά εάν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ενιαίο Μητρώο ή όχι. Επίσης, ένα σύστημα ενημέρωσης για τη θεώρηση που ξεκίνησε το 2015 μπόρεσε να εντοπίσει σφάλματα, παραποιήσεις, αλλοιώσεις ε, σε σφραγίδες εισόδου ή εξόδου και σε σχέση με το θέμα της μετανάστευσης θα ήθελα η Επιτροπή να μας δώσει κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις προοδούς από το Νοέμβριο του 2015 ως προς τον, ε, την οργάνωση των συνοριοφυλακών ε, σε σχέση με τα στοιχεία της Europol που θα έπρεπε για το 2015 να συμπεριλαμβάνουν 215 ακόμη φυλάκια συνόρων και επίσης ποιες είναι οι στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ Europol και Ουκρανίας, αν έχουν ξεκινήσει και αν εξελίσσονται. Για τη μετανάστευση επίσης, δύο ερωτήσεις. Το ποσοστό το ποσοστό απόρριψη θεωρήσεω είναι πολύ χαμηλό, είναι κάτω από το 2%. Παρ' όλα αυτά όμω υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό Ουκρανών ε, πολιτών που παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράνομα, παράτυπα, έχοντας ξεπεράσει τον χρόνο της θεώρησης. Ποιες ε, προτάσεις έχει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι μέτρα μπορεί να προτείνει προκειμένου να ε, εξασφαλιστεί η επιστροφή των πολιτών αυτών της Ουκρανίας. Για το τρίτο ζήτημα, το λαθρεμπόριο βάρος ανθρώπων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες σχέση με τους κινδύνους ένα θέμα πολύ ευαίσθητο, ένα θέμα ευρύτατο. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση από το ανώτατο μέχρι το χαμηλότερο τοπικό επίπεδο. Θα μπορούσαμε όμως να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη επισκόπηση προς τους μηχανισμούς παρακολούθησης όπως αυτοί προβλέπονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τις αρχές της Ουκρανίας και εν τέλει για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Δεν μπορούμε παρά να σημειώσουμε την στράτευση και τις προσπάθειες των αρχών της Ουκρανίας. Ε, πολλά μέτρα ελήφθαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ερωτώ λοιπόν τι είδου δεσμεύσει ακριβώς έχουν αναλυφθεί και έχουν τηρηθεί από τις αρχές της Ουκρανίας. Νομίζω ότι η έκθεση ε, ως προς την καταπολέμηση της διαφθοράς ε, σημειώνει σημαντικές προκλήσεις. Πρέπει να γνωρίζουμε βεβαίως ότι οι αλλαγές σε αυτό το επίπεδο της καταπολέμησης της διαφθοράς, της διαφθοράς απαιτούν πολύ χρόνο. Και ένα γενικότερο ζήτημα που έχω να θέσω σε σχέση με τη μεθοδολογία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εκθέση τη διατυπώνει συστάσει και προτάσει που θα μπορούσαν να περιορίσουν του κινδύνου σχέση με, την, ε, με τι μεταναστευτικέ τάσει και την ασφάλεια. Ε, στο βαθμό που αυτέ οι ε, συστάσεις ωστόσο δεν καταγράφονται στην ενδιάμεση έκθεση, πώς αυτές μπορούν να γνωστοποιηθούν στα κράτη-μέλη και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Πρώτη σειρά λοιπόν ερωτήσεων και κάποια θέματα μπορούν να σας φαίνονται γενικά, αλλά στη λεπτομέρειά τους απαιτούν ε, μια σωστή ενημέρωση για να μπορέσουμε να εξεργαστούμε πλήρω το θέμα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι ευκρινήσει και την ενημέρωση που θα μα προσφέρει. Προ το παρόν περιορίζομαι σε αυτά. Ο σεβασμό των κριτηρίων μπορεί να οδηγήσει σε απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρηση. Είναι κεφαλαίου σημασία εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να διασφαλίσουμε πως τα κριτήρια θα τηρούνται και σε μεταγενέστερο στάδιο. Και όπως είπα εισαγωγικά, τα εξεταζόμενα κριτήρια θα είναι και ο οδηγός για τη συνομοθετική μας διαδικασία και εργασία. Ευχαριστώ όλους τους συντονιστές και οδησηγητές και όλα τα μέλη της Επιτροπής Λίβη για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία ο Πρόεδρος. Πρώτα-πρώτα όμως, καλώς όρισαν οι εκπρόσωποι της ε, Ουκρανίας είναι εκπρόσωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση της χώρας. Πρώτο, να δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή. Και μετά στους συναδέλφους. Κύριε Καγιακό Κασίλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και την εισηγητρία. Ευχαριστούμε για τόσα ερώτησε Όσο αφορά το διάλογο για τις θεωρήσεις, ιδιαίτερα με ξεκίνησε το 2008 και τον Δεκέμβριο κάναμε την ε, τελευταία έκτη έκθεση πρόοδου. Διαπιστώθηκε ότι σημειώθηκε η απαραίτητη πρόεδρος, μεταρρυθμίσεις, δεσμεύσεις, ούτω ώστε να υπάρχει αποτελεσματική και βιώσιμη πρόοδο σύμφωνα με το χαρτί πορεία Επί τη βάση τη αξιολόγηση καταλήξαμε ότι όλα τα κριτήρια πληρούνται σε σχέση ε, με αυτούς τους τέσσερις άξονες του προγράμματος δράσης. Ανακοινώσαμε ότι φέτος θα κατεβάσουμε μια νομοθετική πρόταση ούτω ώστε από το πρώτο να πάει στο δεύτερο παράρτημα η χώρα σε σχέση με τον σχετικό κανονισμό. 12 Απριλίου ε, δημοσιοποίησαμε αυτή μας την ε, ανακοίνωση επίση είπαμε ότι έχει σημειωθεί πρόοδο στη χώρα από την έκτη έκθεση και δόθε, από το Δεκέμβριο δηλαδή. Οπότε έγιναν και άλλα μέτρα στη συνέχεια, υπήρξε συνέχεια στα προϋπάρξαντα μέτρα ούτω ώστε οι μεταρρυθμίσεις να υλοποιηθούν και στην ε, τρίτη σελίδα του σχετικού υπομνήματος μνημονίου έχουμε όλες τις λεπτομέρειες Αυτά υπάρχουν επίση στο γραφό εργασία σε εκείνη την έκθεση που συνοδεύει την πρότασή μας. Επίσης, συνεχίζουμε και παρακολουθούμε την ε, υλοποίηση των έχουν συμφωνήθηκαν για επανεισδοχή και κατάργηση θεώρηση. Αυτά γίνανε στις κοινέ επιτροπές παρακολούθησης και υποπτίας των συμφωνιών. Όλα αυτά τα αξιολογήσαμε και θεωρήσαμε ότι η εφαρμογή προχωράει ικανοποιητικά. όπως και στις άλλες μας ε, στις προηγούμενες συζητήσεις είπαμε ότι όλες αυτές οι ρυθμίσεις αφορούν τα βιομητρικά διαβατήρια. Η Ουκρανία εκδίδει από τις 12 πρώτου του 15 βιομετρικά διαβατήρια σύμφωνα με τα προεπιτούμενα από ΕΚΑΟ και από Ευρωπαϊκή Ένωση και όσον αφορά τα στοιχεία του προσώπου και όσον αφορά τα αποτυπώματα και μέχρι τις 14 του είχαν εκδοθεί ε, πάνω από ένα εκατομμύριο μετρικά διαβατήρια. Πάνω από ένα εκατομμύριο σε κυκλοφορία. Και θα γίνει σιγά σιγά η βαθμία αντικατάσταση όλων των μη βιομετρικών ε, διαβατηρίων. Υπάρχει ως ε, όριο το 2026. Πάντως όποιος Ουκρανός δεν έχει βιομετρικό διαβατήριο πρέπει να υποβαλεί σε θεώρηση διαβατήριο. Αυτά για τα διαβατήρια. Αλλά υπήρξαν και άλλες ερωτήσεις. Ας πούμε κάτι για τα μητρώα, τα μητρώα του πληθυσμού. Είπαμε ότι από 1η Ιανουαρίου θα γίνει αυτή η διασύνδεση των διαφόρων μητρώων. Αλλά και για όλα τα άλλα ερωτήματα της εισηγήτριας θα επανέλθουμε και όλα αυτά θα περιέχονται στην ε, έκθεση που θα ετοιμάσουμε. Ο πρώτος ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Radio Free Europe ήδη έχουν ανέβει κάποιε φωτογραφίε από την συνεδρίασή μα. Για το λόγο, συνάδελφε. Πρόεδρε, συμφωνώ και υποστηρίζω πάσα προσπάθεια για κατάργηση της θεώρηση διαβατηρίου ε, για την ε, Ουκρανία. Ε, για όλα όσα περιέγραψε η Μαρία. Εργάζομαι και στην διακοινωνιστική Επιτροπή συνεργασία με τη χώρα. Ε, Επίση και στην ε, συνεργασία του Κοινοβουλίου με την Βερχόβνα Ράντα, ε, στην Επιτροπή των Διοικητών Μεταρρυθμίσεων και όλα αυτά τα έχουμε συζητήσει. Επίσης, είπαμε για το πώ θα χρησιμοποιήσουμε την νέα ψηφική τεχνολογία, ούτω ώστε η δημόσια διοίκηση τη χώρα να βελτιώσει τι επιδόσεις τη. Πάντως είναι πολύ σημαντικές αυτές οι ρυθμίσεις και τα καινούργια διαβατήρια για θέματα ασφάλειας και διαρρεύση των συνόρων. Και από πολιτικής πλευράς, χωρίς να με γρηγορήσω, είναι σημαντική η πρόοδος αυτή. Γιατί όταν έχουμε σε επαφή με τους Ουκρανούς, μας λένε, καλά, για πέστε μας, ποιο είναι το όφελος για όλα αυτά. Για αυτές τις μεταρρυθμίσεις για το χάρτη πορεία σε σχέση με την ε, σύνδεση τη χώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη μελλοντική ένταξή τη. Αλλά πάντω νομίζω ότι το να πληρούνται όλες οι προποθέσει για την κατάργηση της θεώρηση αυτό θα είναι στοιχείο πολύ σημαντικό για τους ε, Ουκρανούς, θα βελτιώσει το κλίμα στην κοινωνία και θα είναι κάτι το οποίο θα δώσει όθηση και σε άλλες μεταρρυθμίσεις. Δεν ξέρω αν θέλει να ενημερώσω την εισηγήτρια για τη δραστηριότητά μα ε, στα όργανα στα οποία συμμετέχω σε σχέση με την Ουκρανία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπονιλή, ο Πρόεδρο. Άλλο συνάδελφο θέλει το λόγο. Ή το Συμβούλιο, όχι. Λέει η πρόσωπο του Συμβουλίου. κύριε ε, εισηγήτρια θέλετε κάτι να πείτε προς την εκπρόσωπο της Επιτροπής. Απλώς πρώτα να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση που έχει διατυπώσει για την συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωση, ούτως ώστε ε, να προχωρήσουμε για το θέμα, μια που είναι ουσιαστικές οι προσπάθειες και η πρόοδος της ε, χώρας. Οπότε, να λάβουμε υπόψη ότι πληρούνται τώρα τα κριτήρια που έχουμε τάξει και από την άλλη μεριά να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα οποία έχουμε πει για την κάθε περίπτωση κατάργησης ε, θεωρήσεων ότι αυτοί που θα ωφεληθούν περισσότερο για κατάργηση της θεώρησης είναι οι πολίτες της χώρας. Σας ευχαριστούμε. Ασυνήθιστο είναι αυτό το οποίο θα σας αναφέρω, αλλά συνήθως δεν ξεκινάνε δεν είναι ανοιχτέ οι συζητήσει ε, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ σε όλου του συμμετέχοντε, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε και το λόγο στου εκπροσώπου τη Ουκρανική Αντιπροσωπεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν θα θέλετε να πάρετε το λόγο, να κάνετε μια σύντομη παρατήρηση, μια σύντομη δήλωσή σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή και πραγματικά θα είναι πάρα πολύ σύντομη. Σα ευχαριστώ που διοργανώθηκε το θέμα η συνάντηση αυτή τόσο γρήγορα και θα ήθελα να δώσω κάποιες πληροφορίες σε για γιατί είναι τεχνικό το ζήτημα, για τα διαβατήριά μας, όπως αναφέρθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ό,τι αφορά τις ταυτότητες. Από την αρχή του έτους, όλοι οι πολίτες που έχουν λάβει νέα ταυτότητα, ε, έχουν λάβει ταυτότητα που έχει εκδοθεί βάση των νέων βιομετρικών ε, στοιχείων. συνεχίζουμε και τη δουλειά αυτή και συνεχίζουμε να πληρούμε περαιτέρω προποθέσει σε ό,τι αφορά στις 14 Ιουνίου θα, θα, θα υπογράψουμε συμφωνία με την γιατί για την καταπολέμηση του οργανωμένου Κλίματος Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Και λίγο πριν από κάποιες μέρες ο Υφυπουργό ε, της Ουκρανίας για θέματα ε, διαφθοράς ε, παρευρέθηκε στις Βρυξέλλες, συναντήθηκε με εκπροσώπους της Κορεπέρ και δώσαμε λοιπόν κάποιες πληροφορίες και στην κυρία Ισαγητρία για τα επιτεύγματα της Ουκρανίας. Να σας διαβεβαιώσω ότι παραμένουμε εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πρόθυμοι να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση ανακύψει. Γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Και επ' ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ήταν από πάντα το πιο ενθαρρυντικό θεσμικό όργανο σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά και υποστηρίζω και την θέση που ακούστηκε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ουκρανία γιατί το θέμα είναι η μεταρρύθμιση. Λάβαμε ε, διαβεβαίωση της, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πληρούμε πλέον τους όρους και ο κόσμος πρέπει να έχει την αίσθηση ότι ολοκληρώνοντας μια μεταρρύθμιση λαμβάνει κάποιο αντίτιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Ευχαριστώ Λακή πρόεδρος. Το σχέδιο έκθεση θα παρουσιαστεί σε μία από τι μελλοντικές συναντησει τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Θα υπάρχει ευκαιρία συζήτηση και περνάμε λοιπόν περνάμε στα επόμενα τέσσερα σημεία που αποτελούν, συναποτελούν μια κοινή συζήτηση για τη σύνευση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των νήσων Σολομόντων και των ομόσπονδων πολιτείων της Μικρονησίας, του Τούβαλου και Τη δημοκρατία των Ίσων Μάρσαλ για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρηση για διαμονή. Ο κανονισμό 539 του 2009 που αναφέρει τι τρει χώρε ε, που θα πρέπει να έχουν θεώρηση τροποποιήθηκε από τον κανονισμό υπαριθμών 509 του 2014 για τη μεταφορά των χωρών αυτών από το παρατημένο στο παρατημένο 2 και η αναφορά των χωρών αυτών στο παράδειγμα 2 ε, συνοδεύτηκε από μια υποσημείωση η οποία ε, διευκρινίζει ότι η εξαίρεση από το καθεστώς των θεωρήσεων θα ισχύει από την ημερομηνία τη ισχύς της συμφωνίας ε, που θα συναυτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συμφωνίε αυτές θα δώσουν δυνατότητα ταξιδιών χωρί θεωρήσει για του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και για του πολίτε αυτών των τεσσάρων χωρών για μέγιστη περίοδο 90 ημερών σε οποιαδήποτε περίοδο 180 ημερών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ενημερώσει σε ό,τι αφορά την προσωρινή εφαρμογή των συμφωνιών αυτών από την ε, υπογραφή του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνενέσει. Η συγκεκριά μα είναι η κυρία Κάπριλ. Θα ακούσουμε και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα μας παρουσιάσουν αυτή τη συμφωνία για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρηση για βραχή διαμονή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι οι τέσσερι τελευταίε ε, χώρε τη λίστα του καταλόγου των 19. Ξεκινήσαμε πριν από δύο χρόνια με την επεξεργασία του καταλόγου αυτού. Άρα πρέπει να επενέσουμε το έργο αυτό Πρόκειται για μικρέ χώρε αυτέ οι τέσσερι τελευταίε χώρε, αλλά θέλω να τονίσω τη σημασία που έχουν. Γιατί είναι χώρε ΑΚΕ και έχουν προνομιακέ σχέσει. Χάρη στη Συμφωνία του Κοτονού, είναι οι χώρε με τι οποίε η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί πολιτικού διάλογο και πραγματική συνεργασία. Έχει συγκεκριμένε ε, σχέσει και μεταξύ αυτών Είναι ένα θετικό μήνυμα, μήνυμα το οποίο αποστέλουμε. Και προσβλέπω στις πληροφορίες που θα μας δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σαφές ότι σήμερα πλέον ε, οδεύουμε προς την ολοκλήρωση μιας περίοδου η οποία ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια. Θα θέλαμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει γενικές πληροφορίες σε ό,τι αφορά την κατάσταση των μεμονωμένων αυτών χωρών και θα ήθελα να θέσω και ένα ζήτημα το οποίο μου προκάλεσε την προσοχή σε ό,τι αφορά την, ε, το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει μια παράγραφος η οποία αναφέρεται στην περίοδο διαμονής και μιλάμε για τις χώρες που δεν εφαρμόζουν, τις ενώσεις που δεν εφαρμόζουν το Σέγγεν χώρες που δεν συμμετέχουν στον χώρο Σέγγεν αυτές θα έχουν ε, δικαίωμα να παραμείνουν 90 μέρες σε περίοδο 180 ημερών σε οποιοδήποτε από τις χώρες αυτές, ανεξάρτητα από την ε, α, διάρκεια που προβλέπεται για την ε, περιοχή Σέγγεν. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα πει γιατί υπάρχει αυτή η κάπω διαφοροποιημένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά τι χώρες εκτός Σέγγεν. Πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα το οποίο με απασχόλησε λίγο σε σχέση με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα ήθελα να την ευχαριστήσω παράλληλα αυτά για τη συνεργασία τη, Να ευχαριστήσω και του συναδέλφου που με βοήθησαν να προχωρήσουμε γρήγορα το θέμα αυτό και θεωρώ ότι αυτό θα αποβεί προ όφελο των πολιτών των χωρών αυτών. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε, κυρία Γκάμπριελ. Κυρία Καϊ, εγώ θέλετε να λάβετε το λόγο κι εσείς. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ την εισηγητρία όντως. Είναι το τελευταίο κομμάτι από συμφωνία ε, απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Τις εννέα χώρες που ζητούμε να απαλλαγούν από την ε, ε, υποχρέωση θεώρησης, κανονισμός 539. Πρέπει να ολοκληρωθούν λοιπόν διμερείς συμφωνίες απαλλαγής. Τον Οκτώβριο του 2014 το Συμβούλιο απίθυνε οδηγίες στην Επιτροπή για τη διαπραγματεύση των συμφωνιών αυτών. Σε τέλη του 2014 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσει με τις ε, τέσσερις χώρες για τα Ισνήσους, Σολομόντος και το Τούβαλου. Έγιναν οι συνομιλίες στις πρεσβείες τους εδώ στις Βρυξέλλες για τα Μάρσαλ και τη Μικρονησία που δεν έχουν διπλωματικές αποστολές εδώ. Οι συνομιλίες έγιναν με επαφές ε, μέσω αντιπροσωπιών τους και αποστολών τους σε άλλες περιοχές όπως Νέα Υόρκη και ειρηνικό. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι συνομιλίες στα τέλη του 2015 και αρχές του 2016 έγινε η μονογραφή των συμφωνιών. Το κείμενο είναι τυποποιημένο, το κείμενο της συμφωνίας έχει υποβληθεί και στο παρελθόν αντίστοιχο σε άλλες περιπτώσεις στο Κοινοβούλιο και έχει δώσει τη συνένεση του Κοινοβούλιο. Προτείνουμε λοιπόν με τα κείμενα αυτά την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για ε, σύντομη διαμονή μέχρι 90 ημέρες πλην περιπτώσεων ταξιδίου ε, για τον σκοπό της επιτέλεσης επαμοιβή δραστηριότητας. Άρα αυτό δεν, δεν περιβλέπεται για την απαλλαγή από τη θεώρηση. Προβλέπονται οι σχετικοί όροι άρσης της απαλλαγής, ε, δημοσιο συμφέρον, προστασία της δημόσιας ασφάλειας, δημοσιακή υγεία, παράτυπη μετανάστευση επανεισαγωγή απέτηση θεώρηση από ένα εκ των δύο μερών, συμφωνίες με απόλυτη αμοιβαιότητα που ισχύουν και για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως να ταξιδεύουν στις χώρες αυτές. Οι τέσσερις χώρες τώρα που πολύ σωστά επεσήμανε η εισηγήτρια συμμετέχουν στην ε, εταιρική σχέση της ΑΚΕ, Αφρικής Καραβίκης Ειρηνικού, με την οποία έχει πολύ στενή συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως αυτή η αμοιβαία άρση της υποχρέωσης θεώρησης διαβατηρίου θα διευκολύνει πολύ και τις σχέσεις μέσα από την ΑΚΕ με τις χώρες αυτές. Κίνδυνο μεταναστευτικών ροών δεν έχουμε εντοπίσει. καμία ανησυχία δεν έχει εκφραστεί ούτε από υπηρεσία ούτε από κράτος μέλος. Στην τελευταία πενταετία δεν έχουν διατυπωθεί αιτήματα ε, ασύλου, δεν έχουν ε, σημειωθεί περιπτώσεις παράτυπης εισόδου ή παραμονής στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλέπεται προσωρινή εφαρμογή εν ώψη της ε, κύρωσης των συμφωνιών για τον Αγούρου που επίση ήταν κομμάτι αυτή της πρότασης του προτινόμενου καταλόγου. Ο, η τροποποίηση του καταλόγου της θεώρησης το 2014 δεν ε, είδε ανταπόκριση από τη χώρα αυτή και τι εμείς περιλημμένως τους ε, απευθύναμε σχετικά ερωτήματα και άρα γι' αυτό δεν υπάρχει πρόοδος. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Άλλα Κύριε Κυρία Κέντς, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρώτα-πρώτα, ευχαριστίες προς την συνάδελφο Καμπριέλ για το έργο της, για όλα αυτά τα θετικά που είναι για αυτές τις χώρες. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα να έχουμε τη δυνατότητα συνεργασίας χωρίς γραφειοκρατικές δυσκολίες, ώστε να μπορεί να μετακινηθεί ο κόσμος. Και στα πλαίσια της Συμφωνίας ε, Κοτονού ε, και ΑΚΕ. Οπότε, γι' αυτό και θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το πώς θα μπορούμε να έχουμε ε, τέτοιες σημαντικέ αλλαγές ήδη με, στη φάση μετά την Κοτονού κατεβλήθησαν κάποιες προσπάθειες. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κυρία Κέγγε, λέει ο πρόεδρος. Δεν βλέπω κάποιο άλλο δεν θέλει να υποβάλει παρατηρήσει. Σχόλια. Οπότε πάμε και στο επόμενο σημείο τη ημερησία διατάξεω που είναι οι συμβάσει για το ψηφιακό περιεχόμενο. Η κυρία Λαουρίστη είναι η εισηγήτρια. Πρόκειται για νομοθετική πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τέτοιε συμβάσει για προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου. Και όπω είπαμε, για την Επιτροπή μα υπεύθυνη η κυρία Λαουρίστην. Αλλά δεν παρίσταται. Δεν τη βλέπω. Μήπως να περιμένουμε 10 λεπτά. 10 λεπτά την περιμένουμε και μετά θα συνεχίσουμε με την κυρία αλλά ορίστε και τους άλλους και όδης εισηγητές. Διάλειμμα 10 λεπτών. Ladies gentlemen, Και κύριοι, λέει ο Πρόεδρος, να συνεχίσουμε. Η κυρία την ξαναήρθε, οπότε συνεχίζουμε με το σημείο 12 της μερικής διατάξεως. Πρόκειται για την νομοθετική πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τις συμβάσεις ψηφιακού περιεχομένου. Ήδη ε, είπαμε ότι η Λάουρη στην εισηγήτρια και έχει τη σκητάλη να κάνει την εισήγηση και κατόπιν κατά τα συνείδη θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή μας υπέβαλε προς μελέτη αυτό το σχεδίο κειμένου οδηγίας όσον αφορά τις συμβάσεις ψηφιακού περιεχομένου. Πρόκειται για πολύπλοκο έγγραφο. Έτσι θα ρυθμιστεί ε, η χρήση από τους καταναλωτές του ψηφιακού περιεχομένου. Πρόκειται για θέμα της ε, ενιαίας αγοράς. Η ΙΜΚΟ και η ΙΟΡΙ είναι οι κυρίως αρμόδιες επιτροπές δική μας Επιτροπή καλείται όμως να γνωμοδοτήσει λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα προβλήματα για την χρήση και κατανάλωση ψηφιακού περιεχομένου από την φύση τους σχετίζονται με το πρόβλημα της προστασίας των δεδομένων. Κάναμε την πρώτη άτυπη ε, επαφή και αντίστοιχες συνεδριάσεις για το θέμα τούτο. Χθες είχαμε και μια συνάντηση ε, και στον κύριο τράπεζα των συνεισηγητών από τις διάφορες επιτροπές. Ακούσαμε πρόταση για το χρονοδιάγραμμα της εργασίας μας. Δεν αποκρισταλώθηκαν τα πράγματα γιατί δύο επιτροπές δεν συμφώνησαν σε σχέση με το με τι ρυθμό πρέπει να προχωρήσει ε, η δουλειά μας. Επίσης, ε, υπήρχε και το θέμα του κατά πόσο θα έχουμε μία ή δύο εκθέσεις. Γιατί το θέμα είναι ότι κάποια μήλικα αγαθά και υπηρεσίες θα καλυφθούν, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει και άλλη μία για ε, κάποια υλικά αγαθά και υπηρεσίες. Ας πούμε τι γίνεται με τα smartphone. Ε, είπαμε ότι δεν είναι ε, ξεκάθαρο πια από τις δύο εκθέσεις. Αν υπάρξουν δύο θα καλύπτει τα smartphone. Πρόκειται περί ψηφιακού ή είναι απλώς μια συσκευή υλική, χειροπιαστή, ε, πώς κατατάσσεται επομένω. Και εν τούτων προέκυψε το ότι το χρονοδιάγραμμα θα καθοριστεί όταν υπάρξει κάποια συμφωνία σε σχέση με το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Πάντως, σε σχέση με την οδηγία, ελέγχθη ότι είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι το θέμα το τι θα γίνει με την αγορά και πώς είναι δυνατόν να έχουμε αγοραπολισία του ψηφιακού περιεχομένου. Ε, είναι κάτι το ασύνηθες μπορεί κανείς να προβεί σε αγορά καταβάλλοντας το αντίτιμο, εις χρήμα. Αλλά ε, επίσης μπορεί κάποιος να δώσει τα προσωπικά του δεδομένα αντί για πληρωμή. Ε, τι ζητήματα ανακύπτουν, τα οποία είναι περίπλοκα. Πώς δηλαδή να θεωρηθούν τα προσωπικά δεδομένα ε, ως ισοδύναμο Χρήματο. Τι γίνεται με την προστασία τη ιδιωτικότητα σε άλλα ζητήματα. Επίση. υπάρχουν και άλλα ζητήματα για το ότι το ψηφιακό περιεχόμενο δεν είναι κάτι το οποίο καταναλώνεται και τελειώνει. Αλλά μπορεί κανείς να δημιουργήσει νέα δεδομένα Υπάρχουν κάποια άρθρα στην οδηγία ότι με το πέρας της ο καταναλωτής μπορεί να πει ε, πάρτε πίσω ή να μην δώσει το ψηφιακό περιεχόμενο. Αλλά υπάρχουν και όλα τα δεδομένα που γεννήθηκαν κατά τη διαδικασία αυτή. Και όταν γίνεται η χρήση του περιεχομένου, τότε και ο πάροχος έχει πρόσβαση με τα cookies στα προσωπικά δεδομένα του καταναλωτού. Πολλά τα που ανακύπτουν Δυστυχώς ε, στην αιτιολογική έκθεση γίνεται μία μόνο της παλαιάς οδηγίας και όχι σε όλη αυτή τη δέσμη μέτρων για προστασία δεδομένων που ήδη έχει εγκριθεί. Οπότε σας λέω ότι πρέπει πολύ σοβαρά να εργαστούμε, να καταβάλουμε προσπάθεια και η έκθεση αυτή να λάβει υπόψη την δέσμη μέτρων για την προστασία των δεδομένων. Υπάρχουν πολύ σημαντικές διατάξεις στον κανονισμό. Δεν έχει θέματα ορισμών κλπ. Οπότε, νομίζω ότι έχουμε να διδραματίσουμε σοβαρό σπουδαίο ρόλο, ούτως ώστε να υπάρξουν κάποιες διαστάσεις και έτσι το ψυχικό περιεχόμενο να διέβεται από διατάξεις που υπήρχαν σύντονες με την νομοθεσία και προστασία δεδομένων. Να καλύψουμε όλα αυτά τα λεπτά σημεία. Να στο θέμα από τώρα σε δουλειά. Να είμαστε έτοιμοι πριν τις κυρίως αρμόδιες επιτροπές. ούτως ώστε να επηρεάσουν, γιατί εκ των υστέρων δύσκολα κανείς να τις επηρεάσει. Άρα, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε την πρώτη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών για να τα συζητήσουμε. Και στη συνέχεια να έχουμε το σχέδιο της έκθεσης. Μέχρι τις εκτη η έκτου προτείνω και στη συνέχεια να συνεχίσουμε να δώσουμε κάποιες τροπολογίες τον Ιούνιο και έτσι να έχουμε μια πρώτη εκδοχή του κειμένου και να γίνει η ψηφοφορία στην Λίμπε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. έτσι να ληφθούν υπόψη πλήρως των στοχών της κυρίως αρμόδιες επιτροπές. Ας είναι έτοιμοι οι συγητές και οι πολιτικές ομάδες. Θα συμβάλλουμε πάντως, είμαι σίγουρη. και θα μας λάβουν υπόψη άλλες επιτροπές. Ε, ευχαριστούμε κύριε Λαουριστή. Οι σκιώδε ηγητέ τώρα θα λάβουν το λόγο. Μπόνι για το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καταρχάς θα ήθελα να πω ότι είναι χαρά μας να συνεργαζόμαστε με την Μάριο γιατί είναι εξαιρετική συνεργασία και νομίζω ότι στη τελική ανάλυση θα είναι πολύ καλή γνωμοδότηση που θα προετοιμάσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν ε, τις εργασίες για το θέμα αυτό και ε, διαβλέπω διάφορα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν ε, παιδί εφαρμογή τη οδηγία, ορισμό του ψηφιακού περιεχομένου, θα πρέπει να διευκρινιστούν σε όλο το κείμενο. Τι εννοούμε με το ψηφιακό περιεχόμενο και όπω είπε και η Μάριο, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με το ψηφιακό περιεχόμενο και με τις... από συσκευέ. Υπάρχει η σύνδεση με την ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων και υπάρχει και η σύνδεση με τον κανονισμό το γενικό για την προστασία των δεδομένων. Είναι σαφέ λοιπόν ότι χρειάζεται να εξασφαλίζουμε, να εξασφαλίσουμε ότι το κείμενο τη οδηγία δεν θα είναι αντιφατικό ή, εν πάση περιπτώσει, ασύμβατο με το κείμενο του GDPR. Και εδώ ανακύπτουν κάποια ζητήματα. Για τη φορητότητα, η οποία ήδη ρυθμίζεται στο GDPR. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι το θέμα των δεδομένων ως πληρωμή για ανταλλαγή σε ό,τι αφορά υπηρεσίε και προϊόντα. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε σε ό,τι αφορά τη διάσταση αυτή και εκ παραλλήλου θα πρέπει να φροντίσουμε στο σημείο αυτό να μην προβούμε σε υπερβολική ρύθμιση γιατί μπορεί να είναι δύσκολο να διακριθούν τα δεδομένα τα οποία παρέχονται από τον καταναλωτή ως ε, ανταπόδοση από αυτά τα οποία πρέπει να χορηγηθούν προκειμένου να συναυθεί ε, μια σύμβαση ή να εξασφαλιστεί η παροχή της ε, υπηρεσίας. Από την άλλη, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο καταναλωτής και τα δεδομένα, κάθε είδους δεδομένα, θα προστατεύονται σε ό,τι αφορά επίσης το άρθρο 13 και το 16, σε ό,τι αφορά την καταγγελία της σύμβασης. Ένα θέμα σχετίζεται με την ε, ανάκτηση των δεδομένων και των δεδομένων που συνδέονται με τους καταναλωτές. Έχει συζητηθεί το θέμα αυτό. Μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε λοιπόν. Κάποια δεδομένα να θυμόμαστε συνδέονται με στατιστικά στοιχεία σε ό,τι αφορά το προϊόν και την ε, υπηρεσία, όπως για παράδειγμα το πόσο επισκέφτηκαν μία ιστοσελίδα. Θα πρέπει να λαμβάνει ο καταναλωτής ε, πληροφορίες σχετικά με το πόσο φορές επισκέφτηκε και πόσο καιρό έμεινε στην ιστοσελίδα. Αμφιβάλλω, αμφιβάλλω. Αλλά σε ό,τι αφορά για παράδειγμα παιχνίδια, μπορεί να συμμετάσχει ο καταναλωτής με ένα αβατάρ ε, δεν θα άνοιγε αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο, θα μπορούσε ο καταναλωτής να το χρησιμοποιήσει αυτό χωρίς ε, το επιχειρηματικό περιβάλλον. Από την άλλη πρόκειται για μία, αν θέλετε, διεύρυνση της προσωπικότητας του καταναλωτή. Θα πρέπει να την υπόψη αυτό. Και είμαι βέβαιος ότι θα είναι στενή συνεργασία με την Μαριού και με τους άλλους συζητητές προκειμένου να επιλύσουμε και αυτά τα θέματα και όσα άλλα ενδεχομένως ανακύψουν και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε καινοτόμοι γιατί ο τομέα ο ίδιο είναι Σε Ευχαριστώ κύριε Μπόνι, λέει ο πρόεδρο. Τα πάρετε λόγο, το πάρετε λόγο. Κύριε συνάδελφε, σα ευχαριστώ και εξ ονόματο ε, του κυρίου Πίτερσον θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια τα οποία κινούνται και αυτά προ την ίδια κατεύθυνση της εισηγήτριας. Παρά την γοργή ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου υπάρχει ένα τεράστιο χρησιμοποιητό δυναμικό σε ό,τι αφορά τις δυσνοριακές ε, και διαδικτυακές ε, πωλήσει. Ένας λόγος που αποτρέπει τον καταναλωτή είναι ο κατακριματισμός. Γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζουμε την πρόταση να εναρμονιστούν οι κανόνες αυτές, αυτοί σε όλο το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να έχουν τα ίδια δικαιώματα οι καταναλωτές ανεξάρτητα από το που βρίσκονται και από που αγοράζουν από πλευρά της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο προστασίας ε, του καταναλωτή και των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ανάλογη νομοθεσία και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και το θέμα της φορητότητας. Άρα καλό θα ήταν να συζητηθούν οι κανόνες για την καταγγελία συμβάσεων και σε ό,τι αφορά την ανάκτηση των προσωπικών δεδομένων του καταναλωτή και θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ προσωπικών δεδομένων και ανωνυμοποιημένων δεδομένων. Η οδηγία α, θα ισχύει για όλες τις ε, συμβάσεις όπου πληρώνει ο καταναλωτής ή που παρέχει κάποια ανταποδοτική ε, υπηρεσία. Τι σημαίνει το άλλα, οποιαδήποτε άλλα δεδομένα. Και ο κύριος Πέτρης πραγματικά τονίζει ότι προσβλέπει στη συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άλλος κανείς. Όχι. Να. Ρωτήσω αν η κυρία Στάδων Μάρια, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέλει να πάρει το λόγο. Ο κύριος Στάδων Μάρια. Ναι, ευχαριστώ πολύ που δίνετε το λόγο και στην Επιτροπή όντως. Όπως είπε και η συγγετρία είναι πρόταση στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή κοινωνία. Προσπαθούμε λοιπόν να εντοπίσουμε όλα τα προβλήματα, τα κύρια προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει η επιχείρηση, ο καταναλωτής στην προσπάθεια να συμμετάσχει σε μια πραγματική ψηφιακή ενιαία αγορά. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι κανόνες όπως εντοπίσαμε για την ε, διαγραμμική πώληση προϊόντων αλλά και για την διάθεση ψηφιακού περιεχομένου. Τώρα έχουν αρχίσει κάποια κράτη να αρχίσουν, ε, έχουν αρχίσει ήδη κάποια κράτη να τροποποιούν ή να εισάγουν νέα νομοθεσία. Ε, μας λένε δεν θέλουμε να προκύπτουν δεξιά-αριστερά κάποιοι δεσμευτικοί κανόνες ε, που θα εμποδίζουν, μας λένε οι επιχειρηματίες, να διαθέτουμε τα προϊόντα μας στην ενιαία αγορά. Ε, ένα περιβάλλον λοιπόν το οποίο θα είναι προς όφελος των επιχειρήσεων με βάση ένα ενιαίο σύνολο κανόνων για τις επιχείρησεις που θέλουν να πωλήσουν προϊόντα, το ίδιο και για το ψηφιακό περιεχόμενο που θα είναι διαθέσιμο σε ολόκληρη την Ευρώπη και βέβαια συγκρινόμενο ε, αντίστοιχα και με τρίτες χώρες. Οι ανταγωνιστές επίσης θα έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη γιατί θα ξέρουν ότι ε, οι καταναλωτές θα έχουν αντίστοιχα περισσότερη εμπιστοσύνη γιατί θα βλέπουν ότι ισχύουν οι ίδιοι κανόνες παντού. Αυτή είναι η ουσία της πρότασης για τις παρατηρήσεις των Ευρωβουλευτών, κυρίως βέβαια τη θεώρηση της Λίβε αλλά και από άλλες πλευρές, το ευρύ φάσμα που αναφέρατε. Βεβαίως υπάρχουν δύο ιδιαιτερότητες. Κομμάτι μιας νέας διάσταση αυτής της πρότασης που στρέφεται προς το μέλλον αλλά πρέπει να είναι και ασφαλής τεχνολογικά. Ο κύριο Μπόνι ανέφερε ότι υπάρχει ένας ορισμός ευρύτατο του ψηφιακού περιεχομένου. Καλύπτουμε δηλαδή κάθε τύπου ψηφιακό περιεχόμενο ανεξαρτήτως του διάπλου από τον οποίο περνάει η διάθεσή του. Άρα αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει, όπως είπα, ένας ενιαίος, ένα ενιαίο πλέγμα κανόνων. Να μην μπορεί κάποιος από το σχεδιασμό του προϊόντος ή από την επιλογή του διάβλου διάθεσης αυτού να ε, στρεβλώνει την αγορά και να εξασφαλίζει πλεονεκτήματα ή αντίστοιχα κάποιο να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση ανάλογα με το που βρίσκεται στην αγορά. Άρα καλύπτουμε κάθε τύπο ψηφιακού περιεχομένου. Επίσης, την επιλογή αυτή, την ε, κάναμε γιατί είναι τόσο γρήγορες και το γνωρίζετε πολύ καλά οι τεχνολογικές εξελίξεις που πρέπει να έχουμε στη θέση μας κάτι το οποίο θα είναι στεγανό σε σχέση με τις εξελίξεις που έρχονται σύν το χρόνο. Να μην χρειάζεται δηλαδή τροποποίηση σε μερικά χρόνια ε, το νομοθέτημα. Άρα έχουμε όσο το δυνατόν ευρεία περιγραφή του ψηφιακού περιεχομένου για να κλεπτούμε άλλα προϊόντα που μπορεί να προκύψουν στην αγορά σε μερικά χρόνια. Ένα άλλο ζήτημα που θέτει η κυρία Λάρου στην αλλά και άλλη. η προσφορά ψηφιακού περιεχομένου με αντάλλαγμα δεδομένα, κατά κύριο λόγο δεδομένα. Αυτό γιατί είναι όλο και μεγενθυνόμενο κομμάτι της αγοράς. Από την μελέτη αξιολόγηση βλέπουμε ότι τα δεδομένα, και θα σας δώσω αν θέλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες στη συζήτηση, βλέπουμε πάντως ότι υπάρχει ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς και μάλιστα και οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν στο μερίδιο αυτό της αγοράς προβλήματα, γιατί επί παραδείγματι μπορεί να ε, τους παραδοθεί ένα ελαττωματικό προϊόν, αλλά να μην έχουν τη δυνατότητα ε, επιστροφής του ανταλλάγματος το οποίο έχουν προσφέρει ή αποζημίωσης. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι, απλούστατα, η σκέψη ότι δεν υπάρχει λόγος κανείς να έχει λιγότερα δικαιώματα εάν αγοράσει ένα προϊόν δωρεάν το ΣΥΠΗΝ, εντό εισαγωγικών, γιατί καταχωρίζει το όνομά του, την ε, ε, διεύθυνσή του, το ηλεκτρονικό του, την ηλεκτρονική του διεύθυνση, φίλο, ηλικία και ό,τι άλλο στοιχείο μπορεί κανείς να χορηγεί. Και ξέρουμε ότι οι τιμές το 2012 για κάθε διεύθυνση ταχυδρομείου ήταν ε, τουλάχιστον 2 ε, αμερικανικά δολάρια. Λοιπόν, γιατί να το κάνει αυτό, ενώ αν κατεβάσει ένα τραγούδι μπορεί να του κοστίσει 0,99 ευρώ. Λιγότερο δηλαδή, ενώ έχει περισσότερο περιεχόμενο που κτίσει. Γι' αυτό λοιπόν περιλαμβάνουμε και δεδομένα τα οποία προσφέρονται ως αντάλλαγμα για μια αντιπαροχή. Ε, πολλοί ομιλητέ επισημαίνουν το λόγο επί του ΑΕΠ. Προς το παρόν δεν μπορέσαμε να κάνουμε μια αναγωγή σε λόγο ΑΕΠ γιατί δεν είχε υιοθετηθεί η πρόταση, όμω θα διορθωθεί αυτή η έλλειψη. Θα κάνουμε τις αναφορές, τι προσαρμογέ και την αναγωγή σε ΑΕΠ. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να κοιτάξουμε το σκεπτικό πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια. Κοιτάμε το ίδιο θέμα από δύο προοπτικές. Υπάρχει το GDPR, το οποίο κοιτάει το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, απαραίτητο και ευπρόσδεκτο, αλλά από την άλλη έχουμε μία παροχή έναντι αντιπαροχής, ανάλογα με τη φύση της σύμβασης. Και άρα υπάρχει ένα ζήτημα αμοιβέ εξυπηρέτηση συμφυρόντων. Άρα πρέπει η παροχή και η αντιπαροχή να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Εάν υπάρχει ανισορροπία σε αυτό, δηλαδή κάποιο να έχει πληρώσει περισσότερα από την ε, αντιπαροχή που λαμβάνει, τότε προφανώς πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί. Δύο λοιπόν προοπτικές αφενό της ε, προστασίας του ηθικού βίου, αφετέρου της ισότητας σε μια συναλλαγή. Και αυτό προσπαθούμε να επιδιώξουμε, όχι μόνο με την προστασία των δεδομένων στο GDPR, αλλά και την δυνατότητα για τον καταναλωτή που είναι το ίδιο άτομο, εν προκειμένου, να διεκδικήσει τα ενοχικά του δικαιώματα σε περίπτωση που είναι ελαττωματική αντιπαροχή. Πρέπει πάντως να σημειώσουμε ότι μέρη μας ήταν να εφαρμοστεί πλήρως το GDPR. Ήταν απολύτως απαραίτητο να είμαστε βεβαίοι ότι κάθε δικαίωμα του υποκειμένου των δικαιωμάτων θα τηρείται απολύτως. Αυτό διευκρινιστεί σε πολλά ε, σημεία της οδηγίας και ταυτόχρονα. Εάν ο προμηθευτής και επεξεργαστής ε, δεδομένων έχει έντιμη συμπεριφορά σε σχέση με τα δεδομένα θα πρέπει να είναι και σε ε, έντιμη συμπεριφορά του και σε σχέση με την ρήτρα ε, καταγγελία τη ε, σύμβαση. Παραδείγματι, αν καταγγείλω τη σύμβαση για το ελαττωματικό το προϊόν το οποίο μου απεστάλλει, έχω το δικαίωμα, αυτή είναι η πρόταση τη οδηγία, να απαιτήσω από τον προμηθευτή να απόσχει, να, να μην προχωρήσει σε χρήση των δεδομένων μου. Ξεκάθαρα λοιπόν στην οδηγία. Εάν έχει κάνει ένας έμπορος αυτό το οποίο οφείλει δυνάμει του GDPR, δηλαδή αν τα δεδομένα ή τα διαγράψει, τότε έχει καλύψει και τις προϋποθέσεις της οδηγίας. Δεν θέλουμε δηλαδή να δημιουργήσουμε πρόσθετο γραφειοκρατικό φόρτο για τον προμηθευτή, αλλά θέλουμε να τηρηθούν οι διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε απόλυτο βαθμό και επίσης κάτι που ανέφεραν αρκετοί ευρωβουλευτές κατάσταση και επιστροφή της συλλογής δεδομένων σε περίπτωση λύσης της σύμβασης. Θα το πούμε αργότερα βέβαια πιο λεπτομερώς φαντάζομαι, αλλά αυτό το οποίο ουσιαστικά εφαρμόζουμε έχει να κάνει με την υλοποίηση της ε, πάγιας νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όχι μόνο σε επίπεδο ενοχικού δικαίου και προστασία των καταναλωτών, αλλά εν γέννη λέει ότι αν προσφέρονται κάποια δικαιώματα στον καταναλωτή, δεν μπορεί μέσα στην σύμβαση να εισάγονται αντικίνητρα τα οποία θα αποθάρρυναν ή θα εμπόδιζαν τον καταναλωτή από την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Φερρυπίν. Εάν σε μία σύμβαση με την οποία μπορώ να αποθηκεύσω τις φωτογραφίες μου τις οικογενειακές στο νέφος, έχω αποφασίσει να λύσω αυτή τη σύμβαση γιατί δεν με εξυπηρετεί, γιατί δεν είναι ε, σύμφωνη με τα υπεσχημένα. Θέλω να ανακτήσω τις φωτογραφίες μου. Δεν είναι δυνατόν ε, λοιπόν κάποιος να με εμποδίσει, να με μπλοκάρει, να με αποθαρρύνει από την ανάκτηση των φωτογραφιών αυτών και την άρση των δικαιωμάτων μου. Θα τα συζητήσουμε φυσικά αργότερα. Αλλά η βασική ιδέα είναι αυτή και θέλω να υπογραμμίσω πως στόχος μας ήταν να εξασφαλίσουμε πως η προστασία των δικαιωμάτων του GDPR για τους ε, ιδιώτες, για τον ιδιωτικό βίο, πληρούνται απολύτως και ότι δεν επιβάλλει οδηγία, δεν εισάγει οδηγία νέα ε, βάρη και για τον προμηθευτή νέα στην γραφειοκρατική. Αυτή είναι η ιδέα της οδηγίας. Η κυρία Λορεστίν, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή για την συνεργασία και βλέπω ότι υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία θα μπορούσαμε και να σας ξαφνιάσουμε προς τις δύο κατευθύνσεις. Και γιατί ούτε εμείς θέλουμε να επιβάλλουμε πρόσθετους, ε, πρόσθετες επιβαρύνσεις, αλλά και γιατί και εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι ε, εμπόρευμα τα προσωπικά δεδομένα. Και σε αυτό θέλουμε να είμαστε απόλυτα σαφείς και να ορίσουμε αυστηρά όρια. Αλλά ασφαλώς με το διάλογο και τη συνεργασία θα μπορέσουμε να λύσουμε όποια παρεξήγηση ή πρόβλημα. Για μας λοιπόν η λύση θα είναι να περάσουμε μέσα από το κείμενο της προτινόμενης οδηγίας και να συζητήσουμε όλα αυτά τα ευαίσθητα σημεία. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν ε, παρατηρήσεις ή ερωτήσεις, μπορούμε να προχωρήσουμε στις τελικές ε, παρατηρήσεις. Στο τελευταίο σημείο της ημέρας διάταξης, θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας. Η κυρία Κέλλερ είναι η συγκέντρια. Και αυτό ε, κατόπιν της, πρέπει να σημειώσω επίσης ότι κατόπιν της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας η ε, Επιτροπή επέβαλε πρόταση για την τροποποίηση της επαφής του Συμβουλίου του 2015 160 1601 για την υπόθεση της επανεγκατάστασης ε, του το άσυλο από την Ελλάδα και την Ιταλία. Δεν ε, έχει ακόμα οριστεί ο αριθμός των επανακαταστάσεων περί 4.000 ε, προσφύγων. Ε, υπάρχει βέβαια το σχέδιο για την επανακατάσταση Σύρων από την Τουρκία στο πλαίσιο του σχήματος ένας ε, μπαίνει, ένας βγαίνει. Και η κυρία Κέλλερ θα πρέπει να μας μιλήσει για την αλλαγή της νομικής βάσης, αλλά πρώτα θα παρακαλούσα την Επιτροπή να μας παρουσιάσει την έκθεση, την πρόταση. Κύριε Ποσιβέρα και μετά εσείς κυρία Κέλλας. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την πρόταση αυτή. Να σας δώσω το γενικότερο πλαίσιο, όπως και το Σεπτέμβριο, δεδομένη της μαζικής εισρωής μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πρώτη φορά χρησιμοποιήσαμε το άρθρο 38.3 της συνθήκης και εφαρμόσαμε προσωρινά μέτρα προς όφελο της Ελλάδας και της Ιταλίας. 2005 01 είναι το ισχύον νομοθεσία και θα πρέπει να αναθεωρηθεί πλέον. 50.400 από την Ελλάδα, 55.000, 54.000 θα πρέπει να αποφασιστούν σε μετέπειτα χρονική φάση. Το Σεπτέμβριο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταθέσει πρόταση και αν δεν γίνει αυτή η πρόταση, οι 54.000 ε, θα πάνε στην Ελλάδα και στην ε, Ιταλία. Όπως ξέρετε, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη το 2016, τώρα στις αρχές του έτους είχαμε περίπου 2.000-3.000 ε, αφήξεις κάθε μέρα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν να εφαρμόσουν καταπήγοντα μέτρα και στις 17 Μαρτίου αποφασίστηκε στο Συμβούλιο να ε, οριστούν κάποιες αρχές για τη μελλοντική συμφωνία με την Τουρκία υπό τις υφιστάμενες ε, δεσμεύσεις και ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει ενδεχόμενα μέτρα προκειμένου να, επιτρα... να μπορέσει να διευκολυνθεί μια τέτοια συμφωνία, να καταστεί δυνατή. Αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ουσιαστικά τι, να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τους 54.000 που δεν έχουν εκχωρηθεί και να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και πέρα από αυτή, γιατί αυτό που πιστεύουμε είναι το εξή. Επιτρέποντας την είσοδο ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω μιας νόμιμης οδού, ουσιαστικά αποθαρρύνουμε τις παράνομες εισόδους και αυτό θα ωφελήσει τις βασικές χώρες που πλήττονται από την χώρα, την Ελλάδα και την Ιταλία. Προφανώς, όπου ξέρουμε, η κατάσταση στα βορειά σύνορα της Ελλάδας είναι τέτοια που θα πρέπει να υπάρξει ε, ε, αλλαγή των ροών. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε για τους 54.000 αυτούς να χρησιμοποιήσουμε ένα κανόνα λογιστικής ότι τα κρατημέλη έχουν την ευελιξία να πληρούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου μέσω νόμιμης εισαγωγής ενός Σύρου ο οποίος διαμένει στην Τουρκία όχι όμως μόνο επανεκατάστασης γιατί το πεδίο ήταν πιο ευρύ από αυτό που προβλέπεται από τη Συμφωνία 1 προς 1, γιατί το σημαντικό είναι να απαλλαγούν η Ελλάδα, να μειωθούν οι πιέσει στην Ελλάδα και στην Τουρκία και στην Ιταλία και πιστεύουμε ότι αυτό θα επιτευχθεί με πιο πολλέ νόμιμες οδού για είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά και τη συζήτηση που έλαβαν χώρα στα πλαίσια του ΟΗΕ στη διάσκεψη για την εξέβριση τέτοιων νόμιμων οδών για τους μετανάστες δεν ε, συμπεριλάβαμε μόνο την επανεγκατάσταση, αλλά όλα τα νόμιμα μέτρα και τα προγράμματα νόμιμη εισόδου για άτομα τα οποία χρήζουν διεθνού προστασίε. Και πιστεύουμε λοιπόν ότι το κείμενο δεν λέει μόνο και δεν αναφέρει μόνο την επανεγκατάσταση, αλλά όλε τι ε, δυνατότητε ε, νομιμή εισόδου. Θα μπορούσαμε να κάνουμε λοιπόν τροποποιήσεις στην απόφαση του Συμβουλίου, γιατί στην πρώτη απόφαση για την επανεγκατάσταση συμπεριλάβαμε κάποια στοιχεία που δεν λειτουργούν σε ό,τι αφορά την απόφαση του Συμβουλίου. Αλλά ξέρετε ότι είναι συγκεκριμένο το χρονοδιάγραμμα στι αποφάσει του Συμβουλίου και πιστεύαμε ότι πρόκειται για μια πολύ συγκεκριμένη τροποποίηση που είχε συγκεκριμένο σκοπό να δώσει μια ευελιξία στα κρατημέλη σε ό,τι αφορά του μη κορυμμένου 54.000. Δεν θέλαμε να αλλάξουμε του κανόνε όλου εν το μέσο τη διαδικασία. Θέλαμε απλά να δώσουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για τις 54.000 με οποιοδήποτε μέσο. Θα κάνουμε λοιπόν μια πρόταση στο μέλλον για το 54.000 στο μέλλον, αλλά θα αφαιρέσουμε τα άτομα τα οποία έχουν πραγματικά γίνει δεκτά στι επικράτειε των διαφόρων κρατών μελών μέσω των διαφόρων προγραμμάτων. Και γι' αυτό το λόγο ήταν πάρα πολύ σημαντικό να συμπεριληφθεί υποχρέωση στην έκθεση, υποχρέωση κοινοποίηση και έκθεση από πλευρά των κρατών μελών για τα διάφορα πρόγραμματα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μέσω ε, του συστήματος ένας ε, προς ένας ιδιωτικών προγραμμάτων και του καθεξής. Αυτό είναι το πλαίσιο. Είναι πολύ συγκεκριμένη και στόχο θετημένη η πρόταση. Πολύ συγκεκριμένο ο στόχος της και πολύ συγκεκριμένη η κοινωνική βάση. Αυτό είναι το πλαίσιο, είναι πάρα πολύ σύντομη η πρόταση, δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω και φυσικά να, απαντήσω ευχαρίστω στις ερωτήσεις σας. Κυρία Κέλλερ, έχετε το λόγο να παρουσιάσετε και εκθεσή σας. Thank um, Κέλλερ, ευχαριστούμε για την εισήγησή σας. Μίλησαμε για το πλαίσιο που κινούμαστε. Ξέρουμε όλοι πώς έχουν τα πράγματα και δεν συζητήσουμε τώρα τη σημερινή με την Τουρκία, αλλά πάντως προβλήματα υπάρχουν με την πρόταση της Επιτροπής. Να σας τα πω. Πρώτα πρώτα δεν έγινε διαβούλευση με το Κοινοβούλιο. Και όταν είχαμε την πρώτη πρόταση με την κατάσταση, τι κάναμε. Είπαμε άντε αυτή τη φορά να τα καταφέρουμε. Και να μην είναι μόνο διαβούλευση, να έχουμε συνομοθεσία τη δεύτερη φορά. Τώρα όμως πήγαμε στην τρίτη προσπάθεια και πάλι έχουμε διαβούλευση. Αυτό ε, δεν είναι καλό για μας. Οπότε θα πρέπει να αλλάξει, είπαμε, η νομική βάση και να πάμε για συνομοθέτηση. Παρακαλώ να συμφωνήσετε. Αυτά από πλευράς διαδικαστικής και τεχνικής. Τώρα όσον αφορά το περιεχόμενο, ποιο είναι το πρόβλημα. Η πρόταση της Επιτροπής αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Είχαμε την πρώτη απόφαση για την μετεγκατάσταση που έλεγε ότι μετεγκατάσταση πάει να πει μετακίνηση από Ιταλία σε Ελλάδα. Τώρα όμως τους παίρνουμε από εκεί που προβλεπόταν από την Ουγγαρία που έπρεπε υποτίθεται να γίνει η διανομή Ουγγαρία και Ελλάδα και πού θα πάνε. Δεν υπάρχουν πια θέσεις για την ε, με την κατάσταση και συνεχίζουν και ε, φτάνουν ε, άνθρωποι λιγότερο στην Ελλάδα, περισσότερο στην Ιταλία και αυτά μετά τη συμφωνία. Οπότε και αυτοί θα πρέπει κάπου να εγκατασταθούν. Ε, και έχουμε και αύξηση, είπαμε, των αφήξεων σε Ιταλία. Οπότε, α, λύθει ο πρόβλημα της Ιταλίας, τώρα πάμε σε νέους τόπους. Όμως θα πρέπει να ξαναγίνει η μετεγκατάσταση, να είμαστε αλληλέγγυοι προς Ιταλία και Ελλάδα. Τι χρειάζονται την ελληνική ευρωπαϊκή ένωση σε αυτές οι χώρες. Επίσης, αλλάζουμε τελείως το πνεύμα της ε, μετεγκατάστασης όσον αφορά τα πρόσωπα που θα καλύψουμε. Έχουμε την επανένωση των ε, οικογενειών. Αυτό είναι υποχρέωση και τα κρατημέλη. Επίσης ε, άδεια εργασίας. Οπότε δεν έχουμε τη γνωστή ιστορία της επανεγκατάστασης. Και η μετεγκατάσταση ήταν μια απόφαση που υποτίθεται ότι θα αφορούσε 22.000 για κάποιους ευάλωτους από οπουδήποτε. Τώρα όμως περιορίσαμε μόνο ε, τους πρόγραμμους από Τουρκία και τους Σύρους. Και όλοι οι άλλοι αποκλείονται από αυτό το πρόγραμμα της με την κατάσταση. Δεν είναι αυτή η καλύτερη λύση. Έχουμε τον κανόνα του ένας προς ένα που επίσης εκπλήσουν ε, πολλούς ε, τουλάχιστον την πολιτική μα ομάδα, μα δεν νομίζω το κοινοβούλιο κάτι τέτοιο. Θέλει να πάρει κανεί ένα σύρο για να επιστρέψει άλλον έναν. Είπαμε να γίνει σφαιρική προσέγγιση όταν λάβαμε τη σχετική απόφαση για να μην μακρηγορώ. Τι προτείνουμε την έκθεση και αυτά τα έχουμε συζητήσει με τους κοιόδησηγητές ήδη στις συναντήσεις μας. Πρώτα πρώτα να αλλάξει η νομική βάση. Μετά να επαναλάβουμε ότι η μετεγκατάσταση είναι μετεγκατάσταση. Να αξιοποιηθούν οι θέσει για κόσμο από Ιταλία και Ελλάδα. Είναι άλλο πράγμα η επανεγκατάσταση. Αυτά τα, έχουμε πει και τα ξανατονίζουμε στην έκθεση. Τι γίνεται, μεταφέρονται οι θέσει από τον ένα μηχανισμό, μια διαδικασία και πάνε στην άλλη. Αλλά έχουμε και κάποιε άλλες αλλαγέ που θα θέλαμε να επιφέρουμε που νομίζουμε ότι ε, βελτιώνουν την πρόταση. Η μεγαλύτερη ομάδα των μεταναστών είναι οι Αυγανοί. Αυτοί όμως δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα της μετακατάσταση. τουλάχιστον αυτοί προ την Ελλάδα. Ε, Σύριοι, Ιραγινοί και Αυγανοί που δεν καλύπτονται οι Αυγανοί. Και δεν καλύπτονται από αυτό το 185%. Ε, καταλαβαίνω γιατί δεν θέλετε να πειράξετε το κατόφλι και οι περισσότεροι συμφωνούν σε αυτό. Ε, Επίση, στην έκθεση τονίζουμε ότι τα κρατημέλη θα πρέπει να επιταχύνουν τι ενεργέ του και να γίνει η μετεγκατάσταση όσο γίνεται γρηγορότερα. Έτσι θα βοηθηθεί η Ιταλία και η Ελλάδα. Αυτές είναι οι προτάσεις μας. Θεωρούμε ότι έτσι θα αποδώσει η πρόταση αυτή. Θα γίνει το πράγμα γρηγορότερα. Τα συζητήσαμε όλα αυτά τα ζητήματα με τους κοιοδησίγητες και τους ευχαριστώ για τη συνεργασία τους. Και ελπίζω αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί για να ολοκληρώσουμε το έργο μας, το Κοινοβούλιο έστειλε το μήνυμα του και στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν. Θέλουμε να αποδώσει με την κατάσταση. Θέλουμε να προχωρήσει η υπόθεση αυτή γρήγορα. Δεν θέλουμε να είναι μόνο λόγια σύμφωνα με την Τουρκία. Ε, ε, ε, και είπαμε για εκείνη την ανακοίνωση τύπου δηλαδή η μετεγκατάσταση να μετεξελιχθεί, να μεταλλαχθεί σε κάτι τελείως διαφορετικό από το θέλουμε. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Κέλλερ. Μπορούμε να προχωρήσουμε στη συζήτηση τώρα με τους ε, σκιώδεις Με πρώτο, <coughs> τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, We are just waiting for the end of the negotiations. Περιμένω να τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις. Is she there? Is... No, there is no... Okay, just I understood after... Uh, Α, το αντελήφθη εν τέλει ότι δεν είναι εδώ, οπότε θα παρακαλέσω τον κύριο Κύρκο να λάβει το λόγο. Σοσιαλιστές Δημοκράτες. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα μιλήσω ελληνικά και θα σας παρακαλώ να τα ακουστικά σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σχέδιο της για το σχέδιο της έκθεσης και την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε στις δύο συνεδριάσεις των Shadows. Θα ήθελα σε τρία σημεία να σταθώ. Το ένα είναι η αλλαγή της νομικής βάσης και το άρθρο 78.2 ή 78.3. Το άρθρο 78.3 είχε επιλογή είχε επιλεγεί επειδή αναφερόταν σε προσωρινά μέτρα υπέρ των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν επίγουσα κατάσταση λόγω ευνηδίας εισρωής υπηκόων τρίτων χωρών. Η επίγουσα κατάσταση αυτή συνεχίζεται ακόμα. Η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου στην ενημέρωση που μας έκανε σχετικά με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας αλλά και σε ερώτησή μου έκρινε ότι η νομική βάση που προτείνει η Επιτροπή είναι η σωστή. Κατόπιν αυτού και για να μην υπάρχει περαιτέρω εμπλοκή και καθυστέρηση δεν μπορούμε να δεχθούμε την αλλαγή της νομικής βάσης. Δεύτερο, η εισηγήτρια διευρύνει πολύ σωστά το πεδίο εφαρμογή εκτό των Συρίων, Ιρακινών και Ερυθρέων και στου Αφγανού και στην Ελλάδα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό γιατί έχουν εγκλωβιστεί ένας μεγάλος αριθμός Αυγανών οι οποίοι αλλιώ βρίσκονται εντελώς ξεκρέμαστοι. Και βεβαίως αυτό που είπε η κυρία Κέλλερ ότι χάσανε για λίγο, έχουν χάσει και ο αριθμός όμως αυξάνει συνέχεια το threshold, οπότε ίσως έπρεπε να κάνουμε μια εξαίρεση. Ε, το τρίτο, ε, η συγγήτρια θεωρεί ότι 54.000 για την εγκατάσταση πρέπει να παραμείνουν και να χρησιμοποιηθούν 18.000 για την επανεγκατάσταση. Ε, συμφωνούμε απόλυτα. Ήδη υπάρχουν τεράστια προβλήματα με την εφαρμογή τη συμφωνία, γιατί με την κατάσταση δημιουργείται περαιτέρω σύγχυση όταν θέλουμε να συνδυάσουμε αυτού του δύο μηχανισμού. Γι' αυτό συμφωνούμε μαζί τη relocation για relocation, resettlement για resettlement. Άρα, σχετικά με τι τροπολογίε, οι πρώτε 7 που αφορούν την αλλαγή τη νομική βάση δεν γίνονται δεκτέ από εμά. Για τις τροπολογίες 14 και 25 θέλω να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσο τηρείται η για την οικογενειακή επανένωση από τότε που ξεκίνησε η κρίση και με βάση τα στοιχεία και την εμπειρία που υπάρχει μέχρι εδώ, οι δύο εβδομάδες που προτείνει η κυρία Κέλλερ είναι εφικτός χρόνος για να εγκρίνει ένα κράτο μέλος στην μετεγκατάσταση προσφύγων. Αυτά είναι δύο θέματα τα οποία έχουμε ακόμα ανοιχτά. Ήθελα να την ευχαριστήσω για τη συνεργασία της και προσβλέπουμε στην ολοκλήρωση του report με τον καλύτερο τρόπο much, Ευχαριστούμε τον κύριο Κυρκό. Ο κύριος Γιασλόφσκι από το ΙΣΙΑΡ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε λάβει σχετική απόφαση στο παρελθόν και για τη Σουηδία. Φερόταν λοιπόν πως το θέμα που αναλάμβανε η κυρία Κέλλερ θα ήταν πολύ απλό, χωρίς προβλήματα. Συμφωνούσαμε όλοι μεταξύ μας και με την Επιτροπή. Και βλέπω ότι στην ε, υπόθεση όπως ε, τη βλέπουμε πλέον σήμερα, τα πράγματα έχουν περιπλακεί, είναι πολύ πιο περίπλοκα. Θα χρειαστεί συζήτηση επί της ουσίας για την πολιτική που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες η ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών Μεταρρυθμιστών είναι επιφυλακτική και διστακτική έναντι του μηχανισμού επανεκατάστασης που είναι αυθαίρετος, δεν λαμβάνει υπόψη, μετακατάσταση συγγνώμη, δεν λαμβάνει υπόψη το κοινωνικό πλαίσιο και βλέπουμε ότι τα προτινόμενα για την Ιταλία και την Ελλάδα σήμερα κατά κάποιο τρόπο συνιστούν συνέπεια των σφαλμάτων του παρελθόντος. Και δεν θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την πρόταση. Θα θέλαμε να γίνει συζήτηση επί της ουσίας για την πολιτική που θα αναπτυχθεί έναντι των μεταναστών στα επόμενα χρόνια, καθώς οι αποφάσεις για τα 2017-2018 ακόμη δεν έχουν ληφθεί. Αυτά είχα να πω στο στάδιο που βρισκόμαστε. Έχουμε επιφυλάξεις πολύ σημαντικές για το μηχανισμό της μετακατάστασης και δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βιασλόφσκι. Κύριε Νίνα για την άλλη, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστώ ειλικρινά τη Σκά Κέλλερ για την επικοδομητική της προσέγγιση. Μας έδωσε χώρο σε όλους, ήταν πολύ ευχαριστή συνεργασία. Έχω και μια εμπειρία πια γιατί το θέμα επανέρχεται διαρκώς με νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, στο ίδιο θέμα πάντα. Και θέλω να υπογραμμίσω τρία σημεία τα οποία εν μέρη ήδη ε, ανέφεραν οι, δύο συνάδελφοι Θέλω να συμφωνήσω με την προσέγγιση της εισηγήτριας ως προς την ανάγκη να υπογραμμίσουμε πως η νομική βάση δεν είναι η σωστή. Το Σεπτέμβριο του 2015 δεχθήκαμε την ανάγκη για την υιοθέτηση μιας απόφασης του Συμβουλίου με βάση το 38.3 της συνθήκης, καθώς ήταν κατεπίγουσα η ανάγκη και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Από ό,τι φαίνεται όμως ξεκίνησε έτσι ένας παύλος κύκλος και όλα τα, τα επόμενα μέτρα για μετεγκατάσταση ακολούθησαν τη διαδικασία. Η Άλτε θεωρεί ότι αυτό είναι πια υπερβολικό και το Κοινοβούλιο διεκδικεί το ρόλο του συνομοθέτη όπως ορίζεται από τις συνθήκες για το άσυλο και την επικουρική προστασία. Δεύτερον, και πάλι ξεκάθαρα το περιέγραψαν οι συνάδελφοι πριν, η μετεγκατάσταση δεν συνιστά επανεγκατάσταση. Και γι' αυτό η επανεκατάσταση πρέπει να καλυφθεί με επιπλέον ποσοστώσεις, όχι μόνο με αυτές οι οποίες προβλέπονται για τη μετεγκατάσταση, διότι όλοι γνωρίζουμε πως ε, τα νούμερα των ε, μετεγκαθισταμένων είναι τόσο μικρά που δεν μπορούμε να μιλούμε για επιτυχή επιχείρηση ακόμη, τουλάχιστον. Και επίσης ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι α, δεν δουλεύει με, η μετεγκατάσταση, α τη μετατρέψουμε σε κάτι άλλο. Όχι δεν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Πρέπει να εκπληρώσουν τα καθήκοντά του, τα κρατημέλη και τι υποχρεώσει που έχουν αναλάβει. Πρέπει να αναλογιστούμε πολύ προσεκτικά γιατί συνέβη αυτό το. γιατί έχουμε αυτή την αποτυχία. Πρέπει οπωσδήποτε αυτό να μα απασχολήσει και εν ώψη τη αναθεώρηση του κανονισμού που ε, θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Η κυρία Σπινέλη, εκ μέρου τη ΓΚΟΕ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Και πρώτα πρώτα να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια Σκά Κέλλερ για τη δουλειά της που ήταν άριστη όσα έκανε αυτό το σχέδιο κειμένου και για την αποτελεσματική συνεργασία και κυρίως εκτιμήσαμε τα σχετικά με τις διαδικαστικές εγγύσεις Λέει πάρα πολλά για δικαιώματα και εγγύσεις και για το πώς θα γίνει η μετεγκατάσταση και πώς αυτό θα γίνει με συγκεκριμένο και υποχρεωτικό χρονοδιάγραμμα. Επίσης πώς θα έχουμε ε, μια, ένα διαχωρισμό μεταξύ μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης. Είπαμε ότι θέλουμε την αλλαγή της νομικής βάσης. Επ' αυτού επιμένουμε ιδιαίτερα. Είπαμε το άρθρο 78 παράγραφος 2. Αυτό σημαίνει ότι θα συναποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θέλουμε την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου. Στους τελευταίους μήνες το Κοινοβούλιο έχει μείνει απ' έξω από τα όσα εξηφαίνει Συμβούλιο και Επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, αυτό το πρόβλημα. Πρόκειται δηλαδή για αυτού του είδους την ζωή μεταναστών και προσφύγων που δεν έχει προηγούμενο. Έχουμε αυτές τις διακυβερνητικές λύσεις ε, που έχουν χαρακτήρα κατεπήγοντος και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ε, τώρα πια τα, πράγματα δεν γίνονται με τρόπο αυθόρμητο ούτε παραθυρίζουν ότι είναι εξελίξεις ε, οπότε θα πρέπει, όπως λέμε εδώ και καιρό, να βγούμε αυτή τη λογική της λύσης στο γόνατο. Ε, θα πρέπει, εν να εμπλακεί περισσότερο το Κοινοβούλιο ως συνομοθέτης. Αυτό θα πρέπει να διεκδικήσουμε. Εμείς προσωπούμε τους Ευρωπαίους. Να μην γινόμαστε συνένοχοι των αποφάσεων των άλλων πρόκειται για πάρα πολύ εμφυλεγόμενες ε, αποφάσεις. Ακόμα και η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή επικρίθηκε. Δεν ήταν αυτό συμφωνία, αυτό ήταν κάτι σαν δήλωση, statement. Μα έτσι δεν και κανένα είδου κοινοβουλευτικό ε, έλεγχο, κάτι το οποίο επιτάσσει πάσα σύναψη διεθνού συμβάσεω από πλευρά ε, Ευρωπαϊκή Ένωσης και ευχαριστώ ο Πρόεδρος. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Σπινέλη. Άλλα σχόλια. Από τους συναδέλφους του Συμβούλιο, την Επιτροπή. Αν όχι, παρακαλώ την κυρία Κέλλερ να μας κάνει τις τελικές της παρατηρήσεις. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θέλω να ευχαριστώ τους και οδησηγητές για την ευγενή και πολύ καλή συνεργασία. Ε, νομίζω ότι τις προθεσμίες τις έχετε εσείς τώρα, δεν τις έχω πρόχειρες, θα μας τις πείτε. Πρέπει να συντονιστούμε όμως καλά για να απευθύνουμε ένα μήνυμα εύστοχο, καλό και να έχουμε μια καλή τελική έκθεση εν τέλει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Προθεσμία για τις τροπολογίες 9 Ιουνίου 2016, 3 το απόγευμα. 9 Ιουνίου, 3 το απόγευμα. Μια τελευταία παρατήρηση για το θέμα αυτό. Βάσει του άρθρου 39 του κανονισμού έχει διατυπώσει γνωμοδότηση η Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων. Αυτό προβλέπεται σε περίπτωση αλλαγή νομική ε, βάση. Πρέπει λοιπόν το, το αργότερο πριν από την Ολομέλεια, πριν την ψηφοφορία στην Ολομέλεια, να έχει κατατεθεί η γνωμοδότηση νομική επιτροπή. Η πρόταση τη κυρία Κέλλερ για αλλαγή από το άρθρο 78 παράγραφο 3 που ακολουθεί μάλιστα πρόταση, απόφαση του Συμβουλίου κατόπιν νομοδοτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για περίπτωση ευνίδιας ε, εισρωής στο άρθρο 78 παράγραφος 2 ε, και 80 που συνεπάγονται ε, διαδικασία συναπόφασης θα, οδηγεί, θα πρέπει να οδηγήσει μια τέτοια γνωμοδότηση. Φαντάζομαι το γνωρίζει αυτό η κυρία Κέλλερ και είναι διατεθειμένη να ζητήσει στη φάση αυτή της διαδικασίας γνωμοδότηση από την Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων θα συζητήσει ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Νομικών τα θέματα αυτά με τους συντονιστές. Και αν δεν έχετε άλλες παρατηρήσεις, η Επιτροπή παρακαλώ. Μια-δυο πολύ σύντομες παρατηρήσεις. Για την νομική βάση δεν θέλω να επισκεφθώ σε λεπτομέρειες, μόνο υπενθυμίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η Επιτροπή έχει καταθέσει προτάσεις για μόνιμο σύστημα μετεγκατάστασης και για το σύστημα του Δουβλίνου που είναι μακροπρόθεσμη λύση. Εδώ μιλούμε για προσωρινά μέτρα που θα εφαρμόζονται μόνο μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου του 2017. Αυτό φαντάζομαι το γνωρίζετε όλοι. Ήθελα απλώς να σας το υπενθυμίσω εν συντομία. Επίσης, δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η πρόταση να ε, εννοεί ότι μετεγκατάσταση και επανεγκατάσταση είναι κάτι άλλο. Όχι. Άλλο η μετεγκατάσταση, άλλο η επανεγκατάσταση. Απλώς βρίσκουμε ένα μηχανισμό που θα επιτρέψει στην Επιτροπή από πιθανή ποσόστοση κατανομή σε κράτος μέλος να υπολογίσει τον αριθμό των προσφύγων που έχουν μπει στην επικράτειά του. Θα αφαιρεθεί λοιπόν αυτός ο αριθμός των ατόμων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ταυτίζεται η επανεγκατάσταση με την μετεγκατάσταση. Και εν τέλει για να απαντήσω στο σχόλιο του κυρίου Βουλευτή για την επανένωση των οικογενειών. Δεν έχουμε στοιχεία. Είναι πολλές οι περιπτώσεις και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσες υπάγονται στο Δοβλίνο και πόσες είναι με την κατάσταση. Προσπαθούμε να συλλέξουμε τις σχετικές πληροφορίες. Για τη διάρκεια των δύο εβδομάδων, ξέρω ότι στην πρώτη ε, συμφωνία για την ε, μετεγκατάσταση ε, και το ξέρει και η κυρία ε, Κέλλερ είχαμε δώσει ως στόχο δύο εβδομάδες δεν επιτυγχάνεται από τα κράτη-μέλη, από ορισμένα τουλάχιστον, κάποια, όμως, κάποια άλλα όμως προχωρούν πολύ αποτελεσματικά και τα καταφέρνουν. Κυρία Κέλλερ, θέλετε να τίποτα άλλο για να τελειώσουμε. Νομίζω ότι ρωτούσατε την Κομισιόν αν είχε σχόλια, αλλά ακόμη δεν είχε. Δεν ήταν σχόλια αυτά που μας έδωσε. περιπτώσει. Όλα ήταν πολύ ενδιαφέροντα για τις δύο εβδομάδες. Ακριβώς αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ζητούμε ένα μηχανισμό που θα διασφαλίζει την τήρηση αυτής της προθεσμίας. Εάν ένα κράτος μέλος δεν ανταποκρίνεται ε, σε αίτημα των ελληνικών ή ιταλικών αρχών συνεπάγεται ότι έχει δεχθεί τον πρόσφυγα. Και αυτό πρέπει να γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις, πιστεύουμε, αν θέλουμε να επιστρέψουμε έναν μετανάστη και το καθεξής. Νομίζω ότι αυτό θα επιταχύνει πολύ τα πράγματα γιατί έτσι δεν θα βραδιπορεί κανείς στις απαντήσεις του. Ευχαριστώ πολύ τελική νομίζω η δήλωση αυτή της κυρίας Κέλλερ. Κύριε εδώ το πέρα στη συνεδρίαση, η επόμενη στις 30 Μαΐου, την προσοχή Δευτέρα. Τρεις το απόγευμα. Και σας ευχαριστώ.